Good afternoon, ladies and gentlemen. Γεια σας κυρίες και κύριοι. If you want have... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε, λέει ο πρόεδρος. If you want to have your... Ευχαριστώ. Και παρακαλώ να κάνετε ησυχία καθίστε ήσυχα στα καθίσματά σα για να αρχίσουμε ξεκινούμε το, από το παρελθόν ένα σημείο, το οποίο είναι η έγκριση μεσαία διατάξεω, αυτή η οποία σα έχει υποβληθεί, ούτω ώστε να εγκρίνεται το σχέδιό τη ακριβώ όσο έχει τώρα, εάν δεν υπάρχει καμία ένσταση, γιατί έχουμε μόνο ένα σημείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Και αν δεν υπάρχει λοιπόν καμία ένσταση, θεωρούνται ε, εγκριθέντα τα κείμενα τη μεσαία διατάξεω και προχωρούμε στο σημείο αυτό τη μεσαία διατάξεω, όπω σας έχει γνωστοποιηθεί, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του, της 9 η Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των Ρωμά, των Τσιγκάνων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι οι αξιότιμοι συνάδελφοι ε, θα έχουν ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα αυτό με τους αρμοδίους επιτρόπους, την αντιπρόεδρο συγκεκριμένα Vivian Ρέντινγκ, η οποία έχει το χαρτοφυλάκιο για δικαιοσύνη ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, επίτροπο Μάλμστρομ για τις εσωτερικές υποθέσεις αρμόδια και το επιτρόπο Έντερ που έχει την αρμοδιότητα για την κοινωνική πολιτική αλλά επίσης έχουμε και τη συμμετοχή της Επιτροπής Απασχόλησης του Κοινοβουλίου και συμμετέχει στο Προεδρείο της συνεδρίασης και συγκεκριμένα έχουμε εδώ, εξ μου, την κυρία Μπερέ, την πρόεδρο της ε, Επιτροπής που σας είπα. Καλώς ορίσατε. Και επίση, οφείλω να σα υπενθυμίσω ότι απεφάσισε στι 13 Σεπτεμβρίου η διάσκεψη των Προέδρων η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών να διεκπεριώσει αυτήν την παρακολούθηση του θέματο σε σχέση με τι εξελίξει κατόπιν του ψηφίσματο τη 9 Σεπτεμβρίου για του συγκάνου Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Τώρα έχουμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των ε, ε, επιτρόπων που προείπα και συμμετοχή της ε, Task Force που έχει συγκροτηθεί για το ίδιο θέμα. Επίσης είπαμε ότι έχουμε και εκπροσώπους, συναδέλφους της Επιτροπής Απασχόλησης δυνάμει του άρθρου 50 γιατί είναι συναρμόδιοι όσον αφορά την στρατηγική για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ρωμά. Η κυρία Γιαρόκα δε είναι η συντάκτης, η αρμόδια για την έκθεση αυτή. Ήδη έχουμε, έχουμε λάβει υπόψη όλε αυτέ τι μελέτε οι οποίε ε, έχουν ε, γίνει, οι οποίε έχουν διατεθεί σε όλου του αδέλφου που βρίσκονται σήμερα εδώ. Οπότε θα πρέπει να αποδεχθούμε τον κύριο Τζέρομ που είναι ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάρα πολύ σύντομα δε, το Συμβούλιο θα συζητήσει το ζήτημα που ασχολεί σήμερα. Έχουμε δε κάποιες ε, πρωτοβουλίες που έχουν ε, αναλυφθεί, όπως τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την χρήση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση των ε, Ρωμά. Θα γίνει αυτό στο Βουκουρέστι 12 και 13 Οκτωβρίου. Έχουμε πει και μια συνάντηση υψηλού επίπεδου για το ζώμα που την οργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης ή στο Στρασβούργο στις 12 Οκτωβρίου. Πάρα πολύ, σύντομα, όλα, πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά για την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και για την υπόθεση του, της χάρτας του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτως ώστε να έχουμε κάποιες ρυθμίσεις που να είναι νομικά δεσμευτικές. Καλώς ήρθαν και πάλι οι τρεις ε, επίτροποι, αλλά πρώτα θα δώσουμε τη σκητάλη στην ε, κυρία Ρέντινγκ. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει η κυρία Μάλμστρομ και τελευταίος ο κύριος Άντορ. Πάντως θα πρέπει να λεφθεί υπόψη ότι θα δοθεί η ευκαιρία σε πολλούς συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Και προβλέπεται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η συνήθω οταν όταν παρίστανται επιτροπή πρώτα-πρώτα θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές στους οποίους και θα απαντούν οι επίτροποι και κατόπιν οι πολιτικές ομάδες. Και σε τρίτη φάση ατομικά οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές. Όμως σας προτείνω να καταρτιστεί ευθύ εξ αρχής από το δεύτερο γύρο ε, της συζήτησης ε, αυτός ο κατάλογος των όσων να συμμετάσχουν. Και αυτός ο κατάλογος να κλείσει ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα την συζήτηση στα χρονικά όρια που έχουμε. Δύο ώρες. Δύο ώρες περίπου πάμε μέχρι τις 6.30. Επομένω, όποιος θέλει να λάβει το λόγο, να το γνωστοποιήσει στο Προεδρείο, ούτω ώστε να καταρτιστεί και να κλείσει αυτό ο κατάλογο και έτσι να ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτό τον δεύτερο γύρο. Πρώτα-πρώτα. Επομένω. Α, βλέπω, βλέπω. Βλέπω, Όπω προέβλεπα, πρόκειται να είναι μια πολύ ζωντανή συναρπαστική συζήτηση και, όπω έλεγα, θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Α, Περβάνς, μήπως θέλεις να λάβεις το λόγο πριν προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εκ μέρους Επιτροπής των Κοινωνικών Υποθέσεων και εμείς να ευχηθούμε το καλώς όρισες στους επιτρόπους που δέχθηκαν αμέσως την πρόσκλησή μας να έρθουν για αυτήν την ε, συζήτηση που άρχισε τόσο ζωηρά σήμερα το πρωί και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι υπάρχει απήχηση για τα όσα συζητούμε από σήμερα το πρωί. Γιατί και η δική μας ε, Επιτροπή ενδιαφέρεται για αυτή την διαδικασία που έχει αναδευθεί και από τις δύο συνομόνες επιτροπές, ώστε το θέμα για την κατάσταση των συγκάνων να αντιμετωπιστεί και από πλευράς αποφυγής διακρίσεων και από πλευράς ε, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, κατά της φτώχειας. Επομένως, έτσι με αυτό το διτό τρόπο προσεγγίζουμε σήμερα το θέμα και περιμένω πώς και πώς να ακούσουμε θα πούνε οι επίτροποι. Αυτά εισαγωγικά για τη συζήτησή μα και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εγώ ευχαριστώ κύριε Μπερές. Ο κ. και τώρα δίνει τον Πρόεδρο τον λόγο συγγνώμη στην κυρία Ρέντιν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε στι αρχές γενικά ε, αξιολογήσαμε τα πρόσφατα γεγονότα στην Γαλλία και είδαμε το τι ισχύει σε επίπεδο νομικό για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε παρουσιάσεις τις οποίες έκανα εγώ, ο Λάσλο Άντορ και η Σισίλια Μάλστρομ. Καταλήξαμε συλλογικά σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εξής. Το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση του κάθε πολίτη είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαν θεματοφύλακα στη συνθήκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει την πλήρη και ανεμπόδιστη συμμετοχή της από όλα τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για να λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν ε, την δημόσια τάξη και ασφάλεια στο έδαφος του. Κάνοντάς το αυτό θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες οι οποίοι περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2004 για την ελεύθερη διακίνηση να σέβονται τα θεμελιώδη δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και όχι μέτρα τα οποία να βασίζονται στο ανήκειν σε μια συγκεκριμένη εθνότητα. Τρίτον, τελευταίες εξελίξεις στην Γαλλία οδήγησαν σε λεπτομερείς ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Γαλλικές Αρχές για την εφαρμογή του νέου νόμου για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διαβεβαιώσεις τις οποίες έδωσε η Γαλλία σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο στις 22 Σεπτεμβρίου του 2010, ότι δηλαδή, και αναφέρομαι τώρα σε αυτά τα μέτρα και τις διαβεβαιώσεις, ότι τα μέτρα τα οποία έλαβαν οι γαλλικές αρχές το καλοκαίρι δεν είχαν σαν στόχο ή δεν είχαν σαν αποτέλεσμα το να στοχεύσουν μια συγκεκριμένη εθνότητα αλλά καλύπτουν το σύνολο των πολιτών με τον ίδιο τρόπο. Η Γαλλία θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εγκύκλειος της 5ης Αυγούστου δεν ήταν συμβατή με τον συγκεκριμένο προσανατολισμό, αλλά διορθώθηκε και τελικά αντικαταστάθηκε από διαφορετική εγκύκλειος της 13 Σεπτεμβρίου του 2010. Και τέλος, οι γαλλικές αρχές μας διαβεβαίωσαν πλήρως ότι εφαρμόζουν χωρίς καμία διάκριση τις νέες συνθήκες και σύμφωνα πάντα και με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι η Γαλλία επιβεβαιεί την αφοσίωσή της σε μια μορφή στενή συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επαφές με τις γαλλικές αρχές και ήδη σήμερα έστειλε μια επιστολή επίσημη στις γαλλικές αρχές με συγκεκριμένες λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών διαβεβαιώσεων οι οποίες δόθηκαν από πλευρά της Γαλλίας. Τα λόγια καλά είναι, αλλά χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένους κανόνες για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Πέμπτον, για να υπάρξει νομική διαβεβαιότητα σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλους τους πολίτες, των πολιτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτω από δύσκολες συνθήκες, είναι απαραίτητο κάποιες ε, ρήτρε οι οποίες διαδικαστικά περιλαμβάνονται στην οδηγία του 2004 για την ελεύθερη διακίνηση να εφαρμόζονται πλήρως και να μεταφερθούν πλήρως στην ένωμη τάξη των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Γαλλία δεν έχει μεταφέρει την οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση στην εθνική της νομοθεσία. Όχι με τον τρόπο με τον οποίο θα καθιστούσε τις διατάξεις αυτές πλήρως διαφανείς και εφαρμόσιμες. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ότι θα στείλει μια επίσημη προειδοποίηση προς τη Γαλλία ζητώντας την πλήρη μεταφορά στην γαλλική εθνική νομοθεσία της συγκεκριμένης οδηγίας 2004. Εκτός και αν τα μέτρα, τα ενδιάμεσα τα οποία έχουν ληφθεί και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς μας δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, εφόσον πάρουμε περαιτέρω διαβεβαιώσεις από τη γαλλική πλευρά, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε. Αν δεν γίνει αυτό θα αποσταλεί επίσημη προειδοποίηση στα πλαίσια των, του πακέτου διαδικασιών επί παραβάση του μηνός Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει την κατάσταση και σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη στα πλαίσια της οδηγίας για την ελεύθερη διακίνηση για να αξιολογήσει αν θα είναι χρήσιμο να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση εις βάρος και άλλων χωρών. Δεν έχουμε όμως ε, συζητήσει σήμερα άλλα θέματα, άλλες περιπτώσεις. Σήμερα μιλήσαμε μόνο για την περίπτωση της Γαλλίας. Θα μιλήσουμε όμως και για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια των ε, γεγονότων και θα δούμε μεσοπρόθεσμα αν χρειαστεί στα επόμενα πακέτα διαδικασιών επί να στραφούμε και εις βάρος άλλων κρατών μελών για το βασικό θέμα, την κατάσταση των Ρώμα γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε ότι έχουμε μπροστά μας ένα, μια πραγματική κοινωνική και οικονομική πρόκληση και αποτελεί ευθύνη για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη η αντιμετώπιση της. Η ανακοίνωση της 7ης Απριλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαριθμεί μια ολόκληρη σειρά σημαντικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο για να βελτιωθεί η κατάσταση των Ρωμά το ταχύτερο δυνατόν. Προς την κατεύθυνση αυτή και επί τη βάση των εργασιών της πλατφόρμας για τους Ρωμά και της Task Force για τους Ρωμά που ε, δημιουργήθηκε ε, στις 7 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογηθεί η σωστή και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των Ρωμά, θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών στρατηγικών τον Απρίλιο του 2011. Το πλαίσιο αυτό θα βασίζεται στην έκθεση την τελική της Task Force για τους Ρωμά, δεν θα αξιολογεί μόνο τις χρηματοδοτήσεις τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές για την σωστή χρήση των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρωμά. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την καταπολέμηση του αποκλεισμού έχουν θα έλεγα πολυδιάστατες συνέπειες και θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία χαρακτηρίζουν την μειονότητα των Ρωμά. Όλα αυτά θα γίνουν επί τη βάση της ανακοινώσεως για την καταπολέμηση του αποκλεισμού εις βάρος των Ρωμά και της διαδικασίας διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων. Ταυτόχρονα το πλαίσιο αυτό που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει στοιχεία για μια σωστότερη παρακολούθηση και έλεγχο των εθνικών προσπαθειών και στήριξη κυρίως των εθνικών προσπαθειών για τον μη αποκλεισμό των Ρωμά από την κοινωνία. Στα πλαίσια της στρατηγικής ε, του 2020 θα καλέσουμε τα κράτη-μέλη να καταθέσουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ρωμά. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η στρατηγική αυτή στα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα. Θα έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να στηρίξουμε τις λεγόμενες οριζόντιες προοπτικές όπως η ενσωμάτωση των Ρωμά και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει από τα κράτη-μέλη να είναι συγκεκριμένα σε σχέση με τα μέτρα που θα, πάρουν, θα πάρουν στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Θα συνεργαστούμε στενά με όλα τα κράτη-μέλη για την προετοιμασία του συγκεκριμένου πλαισίου για τους Ρωμά και με την υπηρεσία φυσικά ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι θα αναφέρεται τακτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βήματα προόδου που θα έχουν σημειωθεί και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό θα γίνει πριν από το θέρος του 2011. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το, το λόγο στην Επίτροπο Μάλστρομ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα σε υπεύθυνη για θέματα ασφαλεία. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι λειτουργεί η ασφάλεια. Ήταν πολύ δύσκολο να μπω στο κοινοβούλιο. Πολύ αστυνομία υπήρχε εκτό. Τα κατάφερα όμω. Ε, ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους αστυνομικούς γιατί έπρεπε να έρθουμε, αλλά τα καταφέραμε. Δυστυχώς θα πρέπει να φύγω σύντομα. Καταρχήν θα σας δώσω όμως κάποια στοιχεία από τη δική μου σκοπιά. Είναι θαυμάσιο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί τόσο πολύ για το θέμα των Ρωμά και ελπίζω ότι αυτό είναι μια εγγύηση ότι το θέμα δεν θα παραμείνει στα ΜΜΕ μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ότι θα υπάρχει αυτή η έντονη δέσμευση για να βελτιωθεί η κατάσταση τόσων Ευρωπαίων πολιτών. Όπω και εσεί και η ίδια η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική ένδοξη των μειονοτήτων. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμό δεν έχουν θέση στην Ευρώπη. Εκτός από τα νομικά θέματα έχουμε και διάφορες πολιτικές άλλες στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολύψουμε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Παραδείγματο χάρη είναι η οικονομική στήριξη η οποία δίδεται μεταξύ άλλων μέσω των διαφορετικών ταμείων και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Ενσωμάτωσης. το Ευρωπαϊκό αυτό τομείο, υπό μου ευθύνη, γιατί Αυτές οι πολιτικέ πολιτικές βέβαια είναι βασική σημασία στην Ευρώπη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπηκούς τρίτων χωρών και ξέρουμε τους Ρωμά που ζουν στην Ευρώπη δεν είναι υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών αλλά είναι υπήκοοι τρίτου, τρίτου κράτους ή δεν έχουν καμία εθνική υπηκότητα. Η αντιμετώπιση τους βασίζεται στα ίσια δικαιώματα και ευθύνη εναντί όλων των πολιτών που ζουν στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική ένταξη είναι βέβαια μια διτή ε, διαδικασία και από τις δύο πλευρές. Είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και υπάρχει εδώ μοιρασμένη ευθύνη μεταξύ των κυβερνήσεων της Ευρώπης και σε όλα τα επίπεδα η ένταξη αυτή θα πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές, οι τοπικές κυβερνικές οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν το περιβάλλον και τι μπορεί βέλτιστα να πραγματοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ε, κατανομή των βελτίστων πρακτικών. Η, η ένταξη των Ρωμά υπηκότητας τρίτων χωρών μπορούν να γίνουν ε, σύμφωνα με την πολιτική που διαθέτει μέχρι το 2013 850 ε, εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά υπηκός χωρών από διαφορετικά ε, επίπεδα, από διαφορετικές ομάδες, πολιτικές, θρησκευτικέ, εθνοτικές και ούτω καθεξής. Παραδείγματος θα πρέπει να δούμε κατά πόσον τα άτομα αυτά μπορούν να είναι ε, υποψήφια υποψήφια να δεχτούν βοήθεια από το Ταμείο για την ε, χορήγηση ασύλου που διαθέτει 680 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα ταμεία εφαρμόζονται από κοινού, δηλαδή τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για αυτά, για να μην υπάρχει μια διάκριση ανάλογα με την εθνοτική ομάδα στην οποία ανήκουν τα άτομα αυτά. Η μόνη διαφορά που γίνεται είναι αν είναι υπήκοοι ή δεν είναι υπήκοοι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες για συγκεκριμένες δράσεις που εστιάζονται στους, για τους Ρωμά, γιατί αυτές οι πληροφορίες δεν ζητούνται για την προετοιμασία των πολιτών ε, αυτών προγραμμάτων. Όπως ε, προανήκει η Αντιπρόεδρος κυρία Ρέντρινγκ, πολλές φορές στις συζητήσεις μαζί σας, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε μια task force η οποία εργάστηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα. Η ομάδα αυτή θα συνεχίσει να εργάζεται τις επόμενες εβδομάδες για να αξιολογήσει τα διάφορα κοινωτικά ταμεία, τα χρήματα των ταμείων, που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλη του έτους. Και από εκεί και πέρα θα προετοιμάσουμε και ένα ερωτηματολόγιο για να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι τα σχέδια και τα στοιχεία που αφορούν τους Ρωμά υπηκόους τρίτων χωρών στα κράτη-μέλη θα μας δώσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να καθορίσουμε τις πολιτικές μας. Θα ήθελα να σας πω επίσης το επόμενο έτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια ανακοίνωση όσον αφορά την κοινωνική ένταξη υπηκών τρίτων χωρών η ατζέντα αυτή θα συμπεριλαμβάνει κάποιου δείκτε για να υποστηριχθεί αυτή η ένταξη. Παραδείγματο, χάνει εισαγωγικά ε, μαθήματα για τη γλώσσα, η υποστήριξη τη χώρα υποδοχή και ενεργή συμμετοχή των μεταναστών σε όλα τα επίπεδα τη ζωή. Πολλά λοιπόν μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά του υπηκόου τρίτων χωρών. Αυτό είναι η δική μου ευθύνη ο συνάδελφος ε, Επίτροπος Άντερ θα μιλήσει για τα δικά του τα ταμεία που έχει πολλά περισσότερα χρήματα και που μπορεί να συμβάλλουν πολύ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσετε να σας απευθύνω το λόγο και να σας ευχαριστώ για την δέσμευση που έχετε δείξει μέχρι στιγμής και ελπίζω να συνεργαστούμε μακροπρόθεσμα για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτών των πολλών εκατομμυρίων Ευρωπαίων ε, υπηκών. Ευχαριστώ. We pass the floor. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Μάλστον και τώρα ο Επίτροπος Άντερ. Uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, εγώ θα σας μιλήσω για την ε, χρηματοδότηση της ε, κοινωνικής ένταξης. Όμως, πρώτα-πρώτα, Προσεχωγικά να σας πω ότι θέλουμε ε, να έχουμε μια πλατφόρμα κοινών αξιών επί των οποίων έχει τη θεμελιά της Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί όλοι μας αυτά έχουμε αφετηρία, αυτές τις κοινέ αξίες, ό,τι χαρτοφυλάκια και να έχουμε. επίση, θα πρέπει να σας τονίσω ότι είναι ευθύνη της Ένωσης και των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν από κοινού αυτό το πρόβλημα του οποίου ε, η λύση θα εξαρτηθεί από το πόσο θα επιμείνουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, οι τοπικές αρχές, οι διεθνείς φορείς και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και όλοι, όλοι, όλοι. Επίσης, να τονίσω ότι έχουμε αναλάβει δράση για πολύ χρόνο όσον αφορά τη γενική ένταξη των τσιγκάνων. Δεν είναι κάτι το οποίο μόνο από τα πρόσφατα γεγονότα. Έχουμε χράξει τις σχετικές πολιτικές και με συνέπεια προσεγγίζουμε συνεχώ το θέμα και σα παραπέμπω και στην ανακοίνωσή μα τη 7 η Απριλίου όπου όπω προείπε η Αντιπρόεδρος Ρέντιν και συνάδελφο συνάδελφος Μάλμστρομ τόνιζε ότι χρειάζεται μια σφαιρική στρατηγική και προσέγγιση για κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρωμά στην Ευρώπη. Εκεί τάσσονται κάποιε προτεραιότητε δράση για κράτη-μέλη και επιτροπή σε πολλούς Τομεί, σημαντικούς για την υπόθεση τη κοινωνική ένταξης αυτών των ανθρώπων που ξέρουμε ότι έχουν προβλήματα πολλά και αλληλένδετα. Γι' αυτό και έχουμε κάποιες δέκα βασικέ αρχές, γι' αυτή μας την πολιτική, αυτά τα λέει αυτή η ανακοίνωση και έτσι θέλουμε να αναζητήσουμε και να άρουμε τις αιτίε αυτή τη κοινωνική περιθωριοποίηση. και έτσι θέλουμε να έχουμε μέσα πολιτικέ πιο αποτελεσματικά τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών αρχών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών, αλλά και συνεργασία και με τους ίδιους τους Ρώμα. Εκεί επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε προσκολλημένοι ε, και δεσμευμένοι να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της Ένωσης για να πετύχουμε την γενική ένταξη των ανθρώπων αυτών και έχουμε επομένως τα δηλωτικά ταμεία που είναι πάρα πολύ χρήσιμα, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τι εθνικέ προσπάθειε για την βελτίωση τη κατάσταση των Ρωμά. Και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα κρατημέλη ήδη χρησιμοποιούν κοινοτικά κονδύλια για να βοηθήσουν του Ρώμα. Πάντω θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και θα κάνουμε περισσότερα. Πολλέ φορέ μένουν αχρησιμοποιητά τα κοινοτικά χρήματα γιατί χρησιμοποιούνται πάρα πολύ αποτελεσματικά και γι' αυτό και έχουμε προτείνει μια σειρά μέτρων για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Και μεταξύ άλλων είπαμε τον Ιούνιο του 2009 ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί και τροποποιήθηκε ο κανονισμό για το κοινωνικό ταμείο, τόσο ώστε να διευκολυνθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις μέσω του κοινωνικού ταμείου. Και το Περιφερειακό Ταμείο επίσης γνώρισε μια τέτοια τροποποίηση του βασικού του κανονισμού για θέματα στέρασης των ανθρώπων αυτών. Και έτσι μέσω αυτών των κοινοτήτων, με τη συνεργασία, να αξιοποιηθούν περισσότερο τα κοινοτικά χρήματα και σαν αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών διαπιστώσαμε ότι υπάρχει δημιουργικός διάλογος στην Ουγγαρία μεταξύ εθνικών αρχών και των Τσιγκάνων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ θετική αυτή η εξέλιξη, οπότε προχωρήσαμε σε ένα δεύτερο κύμα προσπαθειών στην Ρουμανία τα μέσα Οκτωβρίου. Είχαμε και την συμμετοχή δύο επιτρόπων. Και του χρόνου σε Βουλγαρία και Σλοβακία θα γίνουν παρόμοιε κινήσει. Επίση, όπω έχει δει το Κοινοβούλιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενό πιλωτικού προγράμματο για να έχουμε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια συντονισμού των προσπαθειών για την γενική ένταξη των ε, Ρώμα. Ε, μια προσπάθεια που ξεκίνησε κατά το τρέχον έτος. Τώρα, στις 7 Σεπτεμβρίου αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε αυτή την task force για τους τσιγκάνους. Ε, αυτό το όργανο πρόκειται να αναλύσει και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της, κατόπιν της του Απριλίου. Να διαπιστωθεί πόσο αποτελεσματικά απορροφώνται τα κονδύλια για την υπόθεση της κοινωνικής ένταξης των ε, Ρωμά και θα προσφερθούν τα συμπεράσματα του, της Task Force περί τα τέλη του έτους. μετά προκειμένου να προβούμε σε κάποια ανακοίνωση για το θέμα της αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων και να προχωρήσουμε και σε κάποιες προτάσεις για καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων για το άμεσο μέλλον. Επίσης, μελετούμε το πώς μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών στρατηγικών για Ακριβώς όπως σας τα είπε πριν η κυρία Ρέντιν για να εξασφαλίσουμε πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των προσπάθειων που είναι σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο και έτσι να υπάρχει η αναγκαία υποστήριξη των προσπαθειών αυτών να δούμε τι γίνεται και με τις εθνικές πολιτικές στα εθνικά προγράμματα των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, οπότε να δούμε πώς μπορούμε να τους περιλάβουμε όσον αφορά το, το πρόγραμμα για την Ευρώπη του 2020, για παιδεία, ε, κοινωνική πολιτική κλπ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι μόνο το θέμα του αποκλεισμού της φτώχειας το θέμα του αποκλεισμού ε, της κοινωνικής περιθωριοποίησης, αλλά θα πρέπει συγκεκριμένα στην καινούργια μας ε, πρωτοβουλία και πολύ για την απασχόληση να τους συμπεριλάβουμε και έτσι θα μπορούμε να πετύχουμε κάτι γιατί είναι εξίσου σημαντικό το να δούμε το τι πρόοδος έχει γίνει όσον αφορά την παιδεία και εκπαίδευση ακριβώς όπως ελέγχθηκε και κυρίως για την πρωτοβάθμια παιδεία. Πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να συμμετάσχουν περισσότερο. Όλα αυτά είναι δύσκολα, όλα αυτά είναι προκλήσεις περίπλοκες, τα ξέρετε και θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις δύσκολες από μέρους μας, αλλά αν υπάρχει αγαστή συνεργασία είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε καλά. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρος. Ξεκινάει η συζήτηση συνάδελφοι, διευκρινιστικά. Να πω ότι έχουμε περίπου δύο ώρες μπροστά μας. Και είναι αναμενόμενο ο αριθμός των συναδέλφων που θέλουν να πάρει το λόγο να είναι υψηλότατος. Γύρω στους 25 έχουν ζητήσει το λόγο. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν να προχωρήσουμε είναι να μην ξεπεράσετε παρακαλώ τα δύο λεπτά. έτσι ώστε οι επίτροποι να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα έχουν μια κάποια σημασία να καλωσορίσω και την κυρία Γιαρόκα, την εισηγήτριά μας. Θα της δώσω πρώτη το λόγο και μετά θα προχωρήσουμε στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Και έχει κλείσει ο κατάλογος γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουμε το τάνο 25 μελών που ζήτησαν το λόγο. Κυρία Γιαρόκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφασή της και ελπίζω να οδηγήσει σε τέλος αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Είναι καιρός να καλυφθούν τα νομικά κενά τα οποία υπάρχουν στα κράτη μας, όχι μόνο στη Γαλλία. Υπάρχουν ε, σαν παράδειγμα αποκλεισμοί από την εκπαίδευση, ξεχωριστά συστήματα εκπαιδευτικά κτλ. έχει δίκιο ότι τα μέτρα της ε, γαλλικής κυβέρνησης των γαλλικών αρχών συνιστούν διακρίσεις εις βάρος για λόγους των Ρωμά, για λόγους ε, εθνοτικούς και φιλετικούς. Νομίζω ότι η περίπτωση των Ρωμά έχει πέσει ταυτόχρονα θύμα κάποιων εθνικών εγωισμών και η συζήτηση έχει απομακρυνθεί από τα σημεία στα οποία ε, πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας πώς να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή την φρικτή φτώχεια που χαρακτηρίζει τους Ρωμά και όχι μόνο τους Ρωμά βέβαια σε όλη την Ευρώπη και πώς μπορούμε να δώσουμε ε, μια ευρωπαϊκή ανταπόκριση σε αυτές τις ανάγκες. Να πω ότι τα πολιτικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένα ζητώντας εδώ και έξι χρόνια μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρωμά. Λίγα πράγματα έχουν γίνει και γι' αυτό όχι μόνο σαν Ρωμά αλλά και σαν εισηγήτρια του Κοινοβουλίου εκφράζω τη χαρά μου για το ότι και οι τρεις ε, επίτροποι κάνουν τεράστιες προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι επίσης γιατί βλέπω και αρκετές μεγάλες χώρες να αναφέρονται σε μια κοινή ανάγκη για ευρωπαϊκή απάντηση την προηγούμενη εβδομάδα πριν από την συνάντηση του Συμβουλίου. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή κατετέθη το έγγραφο εργασίας για την ενσωμάτωση των Ρωμά και για τα στρατηγικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν έχουν σημασία οι τίτλοι, οι επικεφαλίδες, αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει ό,τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να δοθεί μια σωστή ευρωπαϊκή απάντηση στα πλαίσια μια σωστή ευρωπαϊκή στρατηγικής για τους Ρωμά. Και ένα τελευταίο θέμα, Πρόεδρε, να πω ότι το βασικό μου επιχείρημα στην έκθεση αυτή ξεπερνά Περνά κάποιες απλές νομικές ρυθμίσεις. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε μια σαφέστατη νομική βάση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ κυρία Γιαρόκα. Διαδικαστικό. Thank you very much, Mr. Chair. I will... Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ήμουν καλή στα μαθηματικά. Αλλά 25 φορές επί ένα λεπτό είναι 25 λεπτά. Και 25 επί 2 είναι 50 λεπτά. 50 λεπτά λοιπόν και δεν καταλαβαίνω, έχουμε τον χρόνο αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Ε, ξαφνικά όταν σήκωσα την κάρτα μου έκλεισε ο κατάλογος των ε, ερωτήσεων και θα ήθελα και εγώ να θέσω μια ερώτηση. Γιατί αλλιώς τι νόημα έχει να είμαι εδώ. Είδαμε εσάς, είδαμε την κυρία Βεζά, είδαμε τον κύριο Μέλος, προσπαθήσαμε να είμαστε δεκτικοί και ευέλικτοι αλλά έχουμε δύο ώρες μόνο μπροστά μας. Θα ακούσουμε τους συντονιστές πρώτα, οι οποίοι θα μιλήσουν για δύο λεπτά ο καθένας και είναι απλά θέμα χρόνου. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, πρέπει να το συζητήσουμε Λοιπόν, έχει κλείσει τώρα πλέον ο κατάλογος, έχετε συμπεριληφθεί στον κατάλογο πλέον και εσείς και οι δύο άλλοι τους οποίους ανέφερα, αλλά σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, οι συντονιστές για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για Κολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι χωρίς καμιά αμφιβολία και οι τρεις επίτροποι που πήραν το λόγο ήλθαν εδώ στο ημικύκλιο για να εκπροσωπήσουν επί της ουσίας τις θέσεις της Επιτροπής και να μας πούνε τι μέτρα θα λάβουν έτσι ώστε να αποκτήσει ένα σαφέστατο ορίζοντα η στρατηγική για τους Ρωμά. Πρέπει να δώσουμε εγγυήσει για την ελευθερία διακίνησης και θα πρέπει να σεβαστούμε την αξιοπρέπεια του ατόμου να διασφαλίσουμε επίσης την ασφάλεια των πολιτών και το θέμα αν θέλετε των Ρωμά είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά γενικότερα και την προστασία των μειονοτήτων. Η Επίτροπος Ρέντινγκ μας είχε πει με ξεκάθαρο τρόπο εδώ και λίγες εβδομάδες πως τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με πιο εύθετο και αποτελεσματικό τρόπο για την βελτίωση των υποδομών που συνδέονται με την ανάπτυξη των Ρωμά. Ίσως κάτι τέτοιο να μην έχει γίνει. Απαιτούνται λοιπόν περισσότεροι έλεγχοι, σκληρότεροι έλεγχοι και ξέρουμε ότι δημιουργήθηκε και από τον Επίτροπο Αντόρ στις 7 Σεπτεμβρίου μια επιτροπή για να συνεργαστεί ε, έτσι ώστε να έχουμε το ταχύτερο δυνατόν νέες συνθήκες για να ξεκινήσει ο διάλογος. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ουσιαστικά και μια διαδικασία προσφυγής επί παραβάση, αλλά το θέμα των Ρώμα είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των κρατών μελών και είναι ένα πρόγραμμα θα έλεγα ιδιαίτερα κοινωνικό. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να μετασχηματίσουμε όπως έλεγε ο Αντόρ αυτό το εμπόδιο σε μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Η εισηγήτριά μας η κυρία Γιαρόκα εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαι πεπισμένος ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να πάρουν μέτρα ξεκινώντας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει μια ρεαλιστική πολιτική γύρω από το θέμα για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ομάδα ο κύριος Μωράης. Δύο είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία είναι υποσυζήτηση σήμερα. Το πρώτο είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει στις πολιτικές ομάδες η κυρία Ρέντινγκ την επόμενη εβδομάδα να συζητηθεί το θέμα αυτό στο σύνολο των Επιτρόπων. Την ευχαριστούμε γι' αυτό και την ευχαριστούμε που το έκανε έγκαιρα. Η προσπάθεια της κυρίας Ρέντινγκ ε, αφορά το θέμα της μεταφοράς της εθνικές νομοθεσίες των διαδικασιών των κοινωνικών και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία επί παραβάση ε, εις βάρος της Γαλλίας ε, για πρώτη φορά θυμίζω γίνεται για παραβίαση μιας βασικής αρχής που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προσπάθεια είναι μια καλή προσπάθεια. Τίθενται ορισμένα ερωτηματικά από πλευρά του κοινού. Η δράση της κυρίας Ρέντινγκ είναι καλοδεχούμενη, αλλά αν σαν παράδειγμα στη Γαλλία είχε υπάρξει μία εγκύκλειος η οποία στόχευε άμεσα τους Ρωμά και ξέρουμε ποια, τι, τι πιστεύει η κυρία Ρέντινγκ γι' αυτό, πώς μπορεί μια τέτοια ρύθμιση να είναι συμβατή με τις ε, αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊκής για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το θέμα δεν είναι μόνο θέμα μη μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία, αλλά είναι θέμα διακρίσεων επίσης ευρύτερα. Επίσης στήθεται το θέμα το ότι έχουμε αγνοήσει τα προβλήματα των Ρωμά, αυτό το ανέφερε και η κυρία Γιαρόκα. Η πολιτική μας ομάδα είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της αναφοράς που θα κάνει τον Απρίλιο μετά την έκθεση της Task Force για τους Ρωμά να μας μιλήσει για την στρατηγική της πολιτικής μας και όχι μόνο για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας να ρωτήσω από την Επίτροπο Ρέντινγκ και από τον Επίτροπο Άντερ. Τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα οδηγούν σε ένα ερώτημα. Καλύτερη χρήση των, κοινωνικών, των κοινοτικών συγγνώμη, κονδυλίων. Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την εκπαίδευση των Ρωμά. Πώς πιστεύετε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν από αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Για την φιλελεύθερη και δημοκρατική ομάδα ο κύριος Αλβάρο. Α, όχι, ο κύριος Αλφάνο, λάθος. Η κυρία Αλφάνο, λοιπόν, ε, με κάθε ειλικρίνεια και σεβόμενος, ε, σεβόμενη αυτά τα οποία ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φοβάμαι ότι γελιοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το να επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, όπως το κάνει στην ανακοίνωσή της, ότι την διαβεβαίωση η Γαλλία ότι δεν ήθελε να χτυπήσει τους Ρωμά, να στοχεύσει τους Ρωμά, ενώ ακριβώς ε, η εγκύκλειος, η υπουργική, η γαλλική, αυτό ακριβώς έλεγε, οδηγούσε ε, σε εκδόσεις, σε απελάσεις, συγγνώμη, των Ρωμά, ειδικά Υπήρχαν και άλλες ε, εγκύκλοι υπουργικές οι οποίες οδηγούσαν σε ένα κυνήγι των Ρωμά. Λοιπόν, δεν θα πρέπει με ένοχο τρόπο να καλύπτουμε αυτές τις αρνητικές ε, ε, ενέργειες. Το να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, το να μην ξεκινήσει άμεσα μάλλον, είναι λάθος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να άμεσα να υπάρξει εκκίνηση της διαδικασίας προσφυγής επί παραβάση Νομίζω ότι είναι σύνηθις η παραβίαση της κοινοτική νομοθεσίας, ιδιαίτερα των οδηγιών που καταπολεμούν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Όλες αυτές είναι παραβιάσεις οι οποίες είναι γνωστές σε όλους. Τις τελευταίες ώρες η Γαλλία θα έλεγα υιοθετεί νέες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι εξίσου, παραβιάζουν εξίσου την κοινοτική οδηγία. Συνιστούν διακρίσεις εις βάρος των Ρώμων και η Γαλλία αυτή τη στιγμή προχωρά σε ε, απελάσεις επί εθνοτικής και φιλετικής αυστηρά βάσεως. Όλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σε σχέση με τον σεβασμό των συνθήκων. Η αδυναμία λοιπόν, η καταστροφική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένη. Η Ιταλική κυβέρνηση κάνει αυτό το οποίο εδώ και χρόνια καταγγέλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα ε, να ε, εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την πρόταση που έχει κάνει ο Μαρόνι και άλλοι της ομάδας του για την υποδοχή των Ρωμά στην Ιταλία. Η κυρία Φλότρο για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Θέλω επί την ευκαιρία να χαιρετήσω την κυρία Ρέντιν και να συνεκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τα σαφή και αυστηρά της λόγια, στο οποίο επέμενε μέσα σε αρκετή πολιτική πίεση. Θα να την ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι αυτό που απόφασισε η Εκτελεστική Επιτροπή σήμερα συλλογικά να αποστείλει δηλαδή μια επίσημη επιστολή που είναι η απαρχή μιας διαδικασίας επί παραβάση. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία για για τις επιπτώσεις τόσο σημαντικές που καταδεικνύουν και άλλες εθνικές νομοθεσίες καταπατήθηκαν ιδίως σας αναφορά για τον ε, μη ατομικό χαρακτήρα της εξέτασης της κατάστασης το θέμα ότι άτομα τα οποία δεν είχαν προειδοποιηθεί και δεν συμφωνούσαν αναγκάστηκαν να δώσουν δακτυλικά από το υπόμετρο κλπ. Και ότι αυτή η εγκύκλωση που εντωμεταξύ ίσως αντικαταστήθηκε αλλά είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Ρωτώμε ε, λοιπόν επ' αυτού τι πρόκειται να κάνει η Κομισιόν όσον αφορά δηλαδή για τις διακρίσεις αυτές και την καταπάμψη των ε, ατομικών ελευθεριών. Τέλος, θα ήθελα ο κύριο Σαντέρ να μας εξηγήσει, γιατί νομίζω θα είναι δύσκολο, όπως το δείχνει η συμπεριφορά της γαλλικής κυβέρνησης ή και της Ιταλικής, γιατί ο κύριος Μαρονή μόλις είπε ότι οι Ευρωπαίοι υπήκοοι χωρίς εργασία θα πρέπει να απελαθούν. Χθες τα είπε αυτά. Αυτό είναι αντίθετο γιατί επί τόπου οι τοπικές αρχές θέλουν να αναπτύξουν συγκεκριμένα προγράμματα για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν και να έχουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για αυτά, γιατί τους μπλοκάρει η κεντρική κυβέρνηση. Πώς θα φροντίσετε λοιπόν εσείς οι τοπικές αυτοδιοίκησεις που το θέλουν να μπορούν παρόλα αυτά να ωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά ε, κονδύλια. Δεν θέλω να σας επενδύσω όλοι ξεπερνάτε τα δύο λεπτά. Άμα συνεχίσουμε έτσι, αποκλείεται να ακούσουμε τις απαντήσεις των επιτρόπων. Ο κύριος Κίχο, πρόεδρε, βέβαια τα κρατημένα θα πρέπει να σεβαστούν την, ελευθερία, την ελεύθερη κυκλοφορία και την νομοθεσία κατά των διακτήσεων και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ακούσαμε την κυρία ε, Ρέντινγκ όσον αφορά τους Γάλλους. Εγώ περιμένω ε, εδώ και αρκετό καιρό να ξέρω ακριβώς τι κάνουν οι Γάλλοι και ποιοι είναι οι νόμοι, ποιοι είναι οι νόμοι που καταπάτησαν. Αλλά με ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπε η κυρία Ρέντιν και όταν αναφέρεστε σε άλλες χώρες συμφωνώ με την προλή σας να έχουμε ένα κατάλογο των ε, χωρών που έχουν επίσης καταπατήσει τα ίδια βασικά δικαιώματα γιατί αυτή τη στιγμή κατηγορούμε μόνο τους Γάλλους θα μπορούσαμε ίσως να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία, να δώσουμε ε, ερωτηματολόγια, να τα πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για να δούμε τι θα γίνει με τις χώρες αυτές τώρα και να μην περιμένουμε κατά πόσον υπάρχουν νέες κατηγορίες για καταπατήσεις. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έγινε με εκείνο το πρόγραμμα που είχαμε σχετικά με τους Ρωμά. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2005 με διάρκεια 10 ετών και συμμετείχαν τουλάχιστον 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε επαρκώς και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η επιτυχία που επιτεύχθη μέσω του προγράμματος αυτού, πράγμα που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι πιστεύουμε στην ποικιλομορφία αντιπολιτιστική πιστεύουμε στην κοινωνική ένταξη, θα πρέπει να σεβόμαστε τους, κανό, τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δίνουμε εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη όσο το δυνατόν γίνεται, ότι θα κάνουν αυτό που θα πρέπει. Γιατί, εν τελευταία αναλύση, τα κράτη-μέλη πρέπει να θεωρούνται ικανά να πάρουν τις σωστές αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των νόμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σταβαρής, εξ Γκουέ. Κύριε Πρόεδρε, για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά το σημαντικό θέμα είναι να μην ξεχαστεί η υπόθεση αυτή. Βεβαίως και απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα, αλλά τα γεγονότα εκείνα τα διαδέθηκαν άλλα, οπότε τώρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και αυτό και θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η υπόθεση που είναι τόσο σημαντική για τις ευρωπαϊκές αξίες να παραμείνει στην επικαιρότητα. Δεν είναι θέμα ελευθερίας διακίνησης, είναι θέμα δυσμενούς διάκρισης ακριβώς όπως είπε ο Κλοντ Μωράης. Θα πρέπει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει. Μια από εδώ πέρα έχουμε μια κατάφορη παραβίαση της σχετικής οδηγίας κατά των δυσμενών ε, διακρίσεων ε, είναι κάτι το οποίο τώρα αποτελεί νόμο ενισχύει και είναι κάτι το οποίο παρεβίασε η γαλλική κυβέρνηση. Επομένως, δεν είναι μόνο θέμα του να κοιτάμε μπροστά και να σβήσουμε το παρελθόν. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να ξέρουμε τι έγινε, ποιος έλαβε τέτοιου είδους μέτρα δυσμενών διακρίσεων. όποιοι έχουν κυκλοφορήσει τέτοια κείμενα θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνε τους. Θα πρέπει να ενεργήσει η ίδια η γαλλική κυβέρνηση και δεν μιλούμε τώρα σε σχέση μόνο με τους ε, Ρωμά. Μιλούμε τώρα για κάτι που αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Αν εκδίδονται, αν απελάβνονται κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλού, αυτό είναι μια μεγάλη κρίση, ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα. Τι γίνεται με την ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Εδώ μιλάμε για κλειδιά εξόδου από την οικονομική κρίση που πούτιθεται εν κινδύνο. Κυρία Ρέντινγκ, ε, μας έκανε υπερήφανος τόσο είπατε πριν από λίγο καιρό. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να, συνεργαστούμε μαζί σας ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις. έτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε και μέσα σε ποια όρια και νομικές ρυθμίσεις την ελεύθερη κυκλοφορία των Ρωμά που ανήκουν στην... των πολιτών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν κανόνες οι κανόνες αυτοί σε πολλές χώρες είναι πολύ αυστηροί και δεν υπάρχει πρόβλημα το να διώχνουν τους νομάδες από τα παράνομα σημεία στα οποία συγκεντρώνονται όπως στην Γαλλία, Ιταλία κτλ. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και στο Λουξεμβούργο σαν παράδειγμα το οποίο το Σεπτέμβριο του 2008 υιοθέτησε πολύ αυστηρούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των νομαδικών πληθυσμών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε με θετικό τρόπο χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία οι οποίες έχουν ουσιαστικά προσαρμοστεί σε αυτή την πρόκληση. Η πρόκληση η οποία έχει θα έλεγα δημιουργηθεί από μια συγκεκριμένη αιτία. Θυμίζω ότι προέρχονται από τη Ρουμανία οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί. Νομίζω ότι τα χρήματα που έδωσαν οι Ευρωπαίοι ε, φορολογούμενοι για την ε, ολοκλήρωση της χώρας αυτής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε επί τη βάση συγκεκριμένων ανηλυμένων υποχρεώσεων από πλευράς της χώρας αυτής. Ενώ τώρα έχουμε να κάνουμε με την βιβλική έξοδο θα έλεγα των Ρωμά από τη Ρωμανία. Να θυμίσω στην κυρία Αλφάνο ότι αυτοί που έφυγαν από τα γαλλικά στρατόπεδα έχουν πάει ουσιαστικά στην Ιταλία και αμέσως προκάλεσαν το ενδιαφέρον των νομαρχιών και στο Τωρίνο και στο Μιλάνο. Ας αποφύγουμε λοιπόν την δημαγωγία για τη συμπεριφορά μιας χώρας η οποία έχει αποδείξει με τη στάση του απέναντι στην σχολική εκπαίδευση των παιδιών των Ρωμά την αφοσίωσή του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται με αυτές τις οργανώσεις οι οποίες ε, ε, υποτίθεται βοηθούν φιλανθρωπικά τους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα πρέπει να μην περνούν υποχρεωτικά τα κονδύλια αυτά από τέτοιες φιλανθρωπικές εισαγωγικά οργανώσεις, αλλά να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Θα ήθελα να ζητήσω από τους επιτρόπους να μην ξεπεράσουν τα δύο λεπτά για να ακούσουμε και τους επόμενους, ε, τρία λεπτά μάλλον, για να περάσουμε και στους επόμενους ε, συναδέλφους που θα θέσουν ερωτήσεις. Πραγματικά θα κάνω ό,τι μπορώ στα δύο λεπτά. Μπορώ πραγματικά να συμφωνήσω με την εισηγήτριά σας. αυτό που είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην αφήσουμε να ξεχαστεί το θέμα, να εργαστούμε κατά της ένδυας. Η Κομισιόν σήμερα ήταν πολύ σαφής. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Δεν θα περιμένουμε αυτού του χρόνου για να δούμε τι θα γίνει. Αυτή η Task Force αναλύει τι γίνεται στις λεπτομέρειες όσον αφορά τα ευρωπαϊκά χρήματα. Η Task Force αυτή θα μας κάνει την παρουσίασή της μέχρι τα τέλη του έτους και από εκεί και πέρα μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα δράσης που προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή με τον συνάδελφο Άνες και τη συνάδελφο Μάρτρομ για τους υπηκούς της ε, τρίτων χωρών. Ο συνάδελφος Άντερ μπορεί να απαντήσει βέβαια. Θεωρώ ότι καλά κατάλαβε το Κοινοβούλιο ότι η απόφαση σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση κατά της Γαλλίας για το τόσο σημαντικό και ουσιαστικό αυτό θέμα που αφορά τα δικαιώματα, τις αξίες της Ένωσης ήταν μία πάρα πολύ ισχυρή χειρονομία. Δηλαδή έχετε όλο το συλλογικό σώμα των επιτρόπων που από κοινού λένε ότι όχι δεν επιτρέπεται να κάνετε αυτά που κάνετε. Γιατί έχουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που δεν έχουν τεθεί στην εθνική νομοθεσία και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ε, προστατευτούν οι πολίτες αυτές σε μια κατάσταση κρίσης. Το άλλο θέμα που δικαίως ετέθη είναι το θέμα των διακρίσεων. Πριν από δύο χρόνια, θυμόσαστε, ξέφερα την απογοήτευσή μου ότι η εγκύκλωση της 5ης Αυγούστου ε, αφορούσε συγκεκριμένα τους Ρωμά. Είπε ξεκάθαρα η Εκτελεστική Επιτροπή αυτό καταπατεί σαφώς την κοινωνική νομοθεσία. Η εγκλήπιος αυτή διορθώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου. Τι έγινε εδώ μεταξύ όμως, μεταξύ της 5 η Αυγούστου και της 13 η Σεπτεμβρίου. Και τι γίνεται σήμερα, αυτή τη στιγμή. Επ' αυτού δεν έχουμε συγκεκριμένε ε, απαντήσεις, συγκεκριμένες αποδείξεις. Η Κομισιόν είναι αναγκασμένη να εργαστεί βάση νομικών αποδεικτικών στοιχείων. Και μπορούσαμε να δράσουμε γιατί είχαμε αυτό το θέμα για την εγκύκλιο. Αλλά δεν είχαμε αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο όσον αφορά το θέμα των διακρίσεων. Λέμε όμως ξεκάθαρα ότι οι διασφαλίσεις που έδωσαν οι γαλλικές αρχές είναι πάρα πολύ θετικές θα πρέπει όμως να δούμε στην πράξη τι γίνεται και γι' αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή έστειλε σήμερα μία επιστολή στην γαλλική κυβέρνηση ζητώντας συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις και συγκεκριμένα θέματα δηλαδή αντίγραφα των ε, διατάξεων απέλασης και και ε, τις διατάξεις για την ε, έξοδο από τη χώρα. Πρέπει δηλαδή να έχουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία, πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας και θέλουμε πολλά, όχι ε, μία και δύο μονάχα, αλλά πολλά για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλυση. Αυτό που είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο είναι ότι δεν είπαμε ότι εντάξει δεχτήκαμε τι μας είπαν οι αρχές και κλείνουμε το φάκελο. Δεν κλείσαμε κανένα φάκελο. Εξακολουθεί να είναι επιτάπητος ο φάκελος και έχουμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου ορίσει στην γαλλική κυβέρνηση για να απαντήσει σε αυτά τα πολύ πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Λεπτομερώς, τι έγινε με τα μεμονωμένα άτομα. Και όταν έχουμε τα στοιχεία αυτά, η νομική υπηρεσία μας θα το εξετάσει και βέβαια θα επανέλθουμε μετά, θα έρθουμε εδώ στο Κοινοβούλιο για να σας πούμε τι έχει γίνει. Ένα τρίτο θέμα που ετέθη είναι τι γίνεται με άλλα κράτη-μέλη βάσει οδηγία ελεύθερη κυκλοφορία. Η Κομισιόν σήμερα εξέτασε την γαλλική περίπτωση. Γιατί εκεί υπήρχε πραγματική πολιτική και κοινωνική διάκριση συγκεκριμένη. Εν μεταξύ όμως η Κομισιόν εξετάζει όλα τα άλλα θέματα της μη εφαρμογής των οδηγιών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία. Πάλι όμως χρειαζόμαστε τα πραγματικά στοιχεία για πραγματική νομική ανάλυση και μόνο όταν κάνουμε αυτό θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια διαδικασία επί παραβάση. Δεν μπορούμε έτσι σφαιρικά να προχωρήσουμε σε διαδικασίες επί παραβάση, γιατί η εφαρμογή της νομοθεσίας σε διάφορα κράτη-μέλη είναι διαφορετική εκάστοτε. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε κατά περίπτωση και να έχουμε μια καλή νομική βάση για να προσάγουμε ένα κράτος μέλος στο δικαστήριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη αλλάζουν την ομοθεσία του, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό νόμο. Εδώ λοιπόν εξετάζουμε αναπερίπτωση και θα αποφασίσουμε και αναπερίπτωση. Υπάρχουν ορισμένε περιπτώσει που μπορούμε να κλείσουμε το θέμα και έχουν λυθεί τα θέματα, τα προβλήματα. Αλλά για τη Γαλλία και αυτή ήταν η μόνη απόφαση που πήρε σήμερα η Κομισιόν. Υπήρχαν οι δύο αποφάσεις αυτές. Η μία να συνεχίσουμε νομική ανάλυση, η δεύτερη να ξεκινήσουμε δικασία του παραβάση. Και ελπίζω να έχουμε αρκετά αποδεικτικά στοιχεία τελικά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση για να μπορέσουμε μία, να καταλήξουμε σε μία νομικά βάσιμη απόφαση. Πάντα υπό την αιγίδα των ε, νομικών μας υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Επίτροπος Άντερ. Focus my ε, intervention on the question what happened. Να σας πω τι γίνεται με τα κονδύλια και τι απορρόφηση σε κάτω μέλος, τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα στο μέλλον. Ας γίνει όμως πρώτα μία διαφοροποίηση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών κράτων μέλος, διότι κάποια από τα παλιότερα κρατημέλη έχουν καταφέρει να συμπεριλάβουν και να εντάξουν την κοινωνία με τη βοήθεια της Ένωσης τους συγκανούς. Όμως υπάρχουν κάποιοι άλλοι όπως η Φιλανδία και η Ισπανία ε, έχουν βέβαια λιγότερους συγκάνους από ότι οι κεντροευρωπαϊκά κράτη ή βαλκανικά κράτη όπου τώρα ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την μεγάλη την πρόκληση. Άρα υπάρχει εμπειρία κτηθήσα από τα παλιότερα κράτη-μέλη ε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν είναι μηχανικά αυτή να τη μεταλαμπαδεύσουμε εκεί, διότι είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα μεγέθη και τα άλλα κρατημέλη τα οποία μπήκαν ε, το 2004. Έχουμε για αυτά τα κράτη μια πενταετή περίπου εμπειρία και γι' αυτό και η Task Force προς τα εκεί θα κινηθεί όσον αφορά τα συμπράσματα τα οποία θα εξαγάγει για την χρήση και απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων να μην βιαστούμε εξαγωγή των συμπερασμάτων. Πρέπει να έχουμε αποτελέσματα κοινωνικά αποτιμητά. Όμως, να λάβουμε υπόψη πάντα τις θετικές εμπειρίες από τις προσπάθειες ε, ένταξης των ε, τσιγκάρων και έχουμε βέβαια το Ίδρυμα Σόρος, την Παγκοσμία Τράπεζα, όλοι αυτοί έχουν βοηθήσει. Οπότε έχουμε ήδη κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε κάποια μέσα ενημέρωση που αφορούν και λειτουργούν με τσιγκάνους και για τους τσιγκάνους, εφαρμός τηλεόρασης, ραδιοφώνου και έχουμε επίση και κάποια προγράμματα που έχουν βοηθήσει τους νεροτσιγκάνους να έχουν προσβασιμότητα στην νοτέρα, τότε παιδεία. Πριν κάτι το, που αυτό δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Οκ, okay, όσον αφορά την στέγαση, ε, εκεί βέβαια υπάρχουν ακόμα προγράμματα, αλλά, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία, θετικά στοιχεία πρόοδου. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε πραγματικά επιτυχίες στους τομείς που προαναφέραμε και στην παιδεία. Εκεί που θα πρέπει να πετύχουμε την αλλαγή είναι το να έχουμε πιο αποδοτικό, καλύτερο τρόπο σχεδιασμού των προγραμμάτων. Δεν μιλούμε μόνο για τους ελέγχους. Βεβαίω και χρειάζονται. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι εκεί ο αδύνατος κρίκος, ούτως είπε. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων πρέπει να αλλάξει. Και ε, δεν είναι το θέμα τα ε, περιφερειακό, το Περιφερειακό Ταμείο, τα Διευθυντικά Ταμεία, αυτά φτιάχτηκαν από πρώτη τριακονταετία, και επομένω δεν σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν για τέτοια δύσκολα πράγματα. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε τις νέες πολιτικές, την πλατφόρμα για το 2020. Και τότε θα μπορούσαμε να ευθυγραμμίσουμε με τις αντίστοιχες πολιτικές την χρηματοδότηση. Σήμερα μόλις μίλησαμε με αντιπρόεδρο της ε, Παγκοσμίου και κάτσαμε και είδαμε τι μπορεί να διερευνηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει γιατί και εκείνη ενδιαφέρεται στο να γίνουν περισσότερα. Περισσότερα και σε συνεργασία με την Ένωση. Το θέμα είναι τι είδους προγράμματα θέλουμε αυτοί να θεωρήσουν ότι είναι θέμα αρμοδιότητας αυτέ οι τράπεζε, αυτοί οι φορεί. εμείς να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να τα πρικοδοτήσουμε αυτά τα προγράμματα. Βέβαια και η συμμετοχή των τοπικών αρχών είναι σημείο κλειδί. Είναι προπόθεση επιτυχία. Και όπως ελέγχθηκε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι κάτι το οποίο απόκειται στα κράτη-μέλη. Του χρόνου και όλε θα είναι νέο κανονισμό για το Κοινωνικό Ταμείο. Και τότε θα διαπιστώσουμε όλα αυτά τα κενά πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, για Βουλγαρία, Ρουμανία, τα πιο πρόσφατα η αλήθεια είναι ότι μπήκαν σε πάρα πολύ δεσμένη οικονομική συγκυρία στην Ένωση. Μπήκανε μέσα στην οικονομική κρίση και έτσι υπήρξε πρόβλημα εκεί χρήση και απορρόφηση των ε, κονδυλίων. Η Ρουμανία έχει χρησιμοποιήσει λιγότερο από το 1% των ε, πόρων που προέρχονται από το κοινωνικό ταμείο. Φυσικά και πρόκειται για την χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Εμείς όμως συνεχίζουμε τη συνεργασία μαζί τους τόσο ώστε αυτού του είδους η διοικητική μελητεία, οι προσπάθειες να βελτιωθούν και έτσι να πάμε σε βήματα πρόοδου. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Είχε κάποια πολύ σοβαρή υποχρέωση η Επίτροπος Μάλμστρομ και έφυγε και άρα τώρα έρθε η ώρα των συναδέλφων. Έχουμε 30 καταγεγραμμένους θα πάμε σε τρεις γύρους ε, συζήτησης ε, περίπου από 10 και για αυτό παρακαλώ μια που είμαστε τόσοι πολλοί να μιλάτε περίπου ένα λεπτό αλλιώς δεν θα προκάνουμε η αξιότιμη κυρία Αντζελίλη έχει το λόγο ούν μινούτο λέει ένα μισή λεπτό μου είπατε. Είμαι πεπισμένη ότι η Επίτροπος Ρέντινγκ θα κάνει τεράστιες προσπάθειες και τις προσπάθειες αυτές θα τις κάνει όχι μόνο για το δικαίωμα για την ελεύθερη κυκλοφορία των Ρωμά και υπερασπιζόμενη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όταν αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζονται με κάπως αφηρημένο τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε όλους τους παρόντες. Πόσοι από εσά πήγατε να επισκεφθείτε ένα, ένα, ένα οικισμό τον Ρωμά το χειμώνα κατά τη διάρκεια μιας βροχερής ημέρας. Να δείτε πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι, πώς ζουν τα παιδιά κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι απλά απάνθρωπες με τα ποντίκια, με τη βρώμα μέσα στα περιτώματα χωρίς καμία, κανένα δικαίωμα. Λοιπόν τώρα τι να μιλάμε για μειονότητα καταρχάς. 12 εκατομμύρια Ρωμά είναι δύο φορές ο πληθυσμός της Ιρλανδίας. Τι μειονότητα, εν πάση περιπτώσει. Και εκνευρίζομαι να χρησιμοποιούμε όλη αυτή τη θεσμική ενέργεια μόνο και μόνο για να κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Ας μην μιλάμε για το παρελθόν, ας μην δυσκολεύουμε τα πράγματα, ας μιλήσουμε για μια στρατηγική ιδιαίτερα για τους ανηλίκους Ρωμά. Γιατί αν δεν υπάρξει διαβεβαίωση του δικαιώματος στην παιδεία των νέων Ρωμά, δεν θα υπάρξει μέλλον γενικότερα για τους Ρωμά. Τελευταία παρατήρηση ε, για τον άλλο επίτροπο. Μη μου μιλάτε για τη Φιλανδία, γιατί δεν είναι σοβαρή υπόθεση. Ας μιλάμε για σοβαρά πράγματα και ας μην μεταφέρουμε τις ευθύνες στις τοπικές αρχές, γιατί οι ευθύνες ανήκουν σε όλους και θα πρέπει να ανοίξουμε μια νέα σελίδα. Ε, κοιτάξτε, επιμένω, αν ο καθένας από εσά παραβιάζει το χρόνο που έχει στη διάθεσή δεν προλάβουμε. Από εδώ και πέρα παρακαλώ όλες οι παρεμβάσεις που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και έγκυρες, αλλά προσπαθείτε να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια πράγματα, ας μην επαναλαμβάνετε τι τις ίδιες παρατηρήσεις, ας κάνετε νέες προτάσεις και να μην ξεπερνάτε το ένα λεπτό καθένας. Τώρα, η Επιτροπή... Köszönöm a Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την καλή τύχη για δύο λόγους. Πρώτον γιατί εδώ και τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατέληξε σε μια θέση ευρωπαϊκή για τους Ρωμά και δεύτερον γιατί η Επιτροπή Απασχόλησης υιοθέτησε μια έκθεση για την ενσωμάτωση των Ρωμά ήδη από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη είναι να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στη σχολική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση γενικότερα και στην απασχόληση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά το Περιφερειακό Ταμείο, το Κοινωνικό Ταμείο να αξιολογήσουμε σωστά επίσης τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και να αξιολογήσουμε επίσης την αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των μέσων. Ορίστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συνοπτική. Νομίζω ότι για το χρονοδιάγραμμα η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον μήνα Απρίλιο είχε πολύ μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε τώρα να την εφαρμόσουμε σωστά η φτώχεια μερικές φορές περιορίζεται θα έλεγα σε συγκεκριμένες μικροπεριφέρειες. Γι' αυτό τα προγράμματα αυτά στα οποία θα καταλήξουμε θα πρέπει να στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών όλων αυτών των μικροπεριοχών. Τα χρήματα λοιπόν δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιηθούν σωστά, αλλιώς δεν θα υπάρξει ελπίδα. Πρέπει να βοηθηθούν οι Ρωμά και στις βιοτεχνικές τους δραστηριότητες να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε οικονομικά, να τους δανειοδοτήσουμε γιατί δεν μπορούν να δανείζονται από τις τράπεζες, να διασφαλίσουμε σωστές συνθήκες ενσωμάτωσής τους κοινωνικής. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα ή ότι δεν δαπανώνται σωστά τα χρήματα αυτά, αλλά το ότι η κρίση έχει ε, μειώσει το σύνολο των χρημάτων αυτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο και σε ένα λεπτάκι πρώτα πρώτα να συγχαρώ την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ. Μας τα είπε ξεκάθαρα, μας τα είπε αποτελεσματικά για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Υπενθυμίζω ότι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ένας από τους νεοτηρισμούς της συνθήκης της Λισαφώνας και που έχει πλέον δεσμευτική ισχύ. Όμως θέλουμε να καταπολεμήσουμε ε, τις δυσμενείς διακρίσεις. Θέλουμε να υπάρχει πραγματική στην πράξη ελευθερία διακίνησης. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεσμές διακρίσεις βάρος των τσιγκάνων και να μένουν ατιμόρυτες. Και οι τσιγκάνοι και οι αρχές υπόκεινται στους νόμους. Αυτό θα πρέπει να γίνει πράξη ακριβώς αυτό το οποίο είπε η Επίτροπος Μάλμστρομ όταν αναφέρθηκε στο ότι δεν θα πρέπει μόλις περάσει από την φρέσκια επικαιρότητα το ότι έγινε να ξεχαστεί και να δώσουμε μόνο μάχη για την αποτελεσματική ένταξη την κοινωνική των ανθρώπων αυτών. Πρόεδρος, κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ πάρα πολύ σύντομη. Καταρχήν θα ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ. Θέλω να το πω παρόλο που θα μου πάρει από το χρόνο μου. Δεύτερον, έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που αναφέρεται στις 15 Οκτωβρίου. Ας πούμε ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν θα κάνει τίποτα. Τι θα γίνει, ποια είναι η περαιτέρω διαδικασία και τι θα σημαίνει αυτό για τους Ρώμα. Από την άλλη μεριά, αν θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει πραγματικά κάποια αλλαγή και η αλλαγή τη οδηγία θα γίνει όπως πρέπει. Αυτό τι θα σημαίνει για τους Ρώμα που έχουν ήδη απελαθεί. Αυτό θέλω να μου πείτε. Και δεύτερον, η task force αυτή θα πρέπει να δράσει όχι μόνο για την Γαλλία αλλά και γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Και καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι εμείς εδώ ως βουλευτές θέλουμε να εμπλακούμε και όχι μόνο με ανακοινώσει, αλλά μας κάνετε μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκμεταλλευτώ το χρόνο μου. Καταρχήν, πόσο ρεαλιστικό είναι ότι τα ε, κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από την Κομισιόν όταν θα πρέπει να εξοικονομήσουν τα ίδια ακόμα και εν ώψη το ότι η ε, σωμάτωση εκείνων που ε, ζουν εδώ και πολλά χρόνια στις χώρες αυτές έχει λειτουργήσει εδώ 30-40 χρόνια ιδίω μια που φαίνεται στην Ευρώπη έχουμε μια εξέλιξη ε, κατά την οποία φαίνεται υπάρχει μια επιστροφή στις εθνικές αν θέλετε ρίζες βλέπουμε ε, είμαστε κατά των διακρίσεων, κατά του ρατσισμού, έχουμε διαρθρωτικά ταμεία, ταμεία ε, κοινωνική ένταξη κλπ. Όλα αυτά μου φαίνονται πάρα πολύ πολύπλοκα. Δεν άκουσα κανένα που να ε, του αρέσει να υποβάλει αιτήσει σε τόσο πολύπλοκε καταστάσει Και τέλο. εάν έχουμε μια οδηγία από το 2004 θα έπρεπε αυτή το αργότατα να έχει εφαρμοστεί μέχρι το 2006 Μήπως εδώ έχουμε μια καθυστέρηση εφαρμογής γενικά στα κράτη-μέλη που πρέπει να έχουμε καλύτερα κατά νου. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο. Ε, κύριε Επίτροπε, όχι δεν πρέπει να μιλούμε μόνο για ελεύθερη διακίνηση και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εδώ είχαμε και εξατομικευμένη αντιμετώπιση Επίση η κοινότητα των ε, τσιγκάνων έχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω τη. Ε, λάβετε το αυτό υπόψη και όσον αφορά τι διευρύνσει, γιατί τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε θέμα τη ίδια τη δική μα ιστορία. Έχουμε το ότι σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τελούσαν υπό δουλεία οι άνθρωποι αυτοί. Και μιλάμε για χώρε που τώρα πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τώρα σε ε, κάποιες χώρες Ανατολικής Ευρώπης που έχουν δώσει ηθαγένεια. Ε, ολόκληρη η ιστορία έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για το πώς αυτοί οι διοκόμενοι ζητούσαν ε, εδώ και εκεί ε, καταφύγιο. Το εν τρίτον των ε, τσιγκάνων ούτε καν ξέρουν ή δεν ελπίζουν ότι ποτέ θα μάθουν τα δικαιώματά τους. Επομένω, θα πρέπει να του αντιμετωπίσουμε, να του βλέπουμε σαν μέλλοντε εν δυνάμει πολλή Ευρωπαϊκή Ένωση του ανθρώπου αυτού. Ο επόμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επί τη ουσία συμφωνώ 100% τα όσα είπε ο κύριο Κοέλιο και στο λεφτό για να συγκονομήσουμε χρόνο τώρα και επί, επί, του τύπου, επί, του ύφου. Εδώ, εδώ, εδώ είμαι κύριε Ρεντίν. Εάν κατάλαβα καλά, πρόκειται να ε, στείλετε επιστολή προς την Γαλλική Δημοκρατία και μέχρι τις 15 Δεκάτου είπατε ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ανελευθεί κάποια ενέργεια. Εάν επομένως το τόσο όλα τα στοιχεία η Γαλλία δεν θα ανελευθεί καμία ενέργεια. Παρακαλώ απαντήστε μου σε αυτήν την ερώτηση με ένα ναι ή με ένα όχι και δεν θα προβείτε σε αγωγή επί παραβάση. Ε, θα ήθελα αυτό να εξηγηθεί γιατί Αυτά που τα συζητάμε τώρα για του συγκάνου, αυτά μπορεί να γίνουν σε, για, για οποιονδήποτε. Τι κάνει η Κομισιόν. Βλέπω εδώ σε αυτό το νομικό φυλάδιο ότι η μεταφορά της ε, οδηγίας στο ιστορικό δίκαιο ε, προϋπέθεται κάποια έγγραφα τα οποία διαβίβασε η Γαλλία ή στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 και το 2007 τρει διαφορετικά κείμενα τα οποία αφορούσαν την εφαρμογή της οδηγίας μετά τη μεταφράση του ιστορικού Έγινε αυτό Εσεί όμω δεν κάνετε τίποτα. Μισό αυτό κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι κάτι αυτό το οποίο ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό γίνεται στη Γαλλία, αλλά ε, του αφορά όλου. Επομένω, μεταξύ 2007 και 2010 δεν έλαβε ενέργεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έναντι τη ε, Γαλλία. Και τώρα μα εξηγεί η Κομισιόν ότι τελικά έγινε κακή εφαρμογή τη οδηγία, κακή μεταφορά τη οδηγία. Ωραία, τι έγινε, γιατί δεν έγινε τίποτα. Βεβαίω και έγινε κακή μεταφορά. Και Πέστε μας γιατί δεν κάνατε τίποτα, γιατί δεν έλαβαν ενέργειες οι υπηρεσίες σας. Η τελευταία, η... εσείς κυρία μου για αυτό το γύρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω ικανοποίηση όσον αφορά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ξεκάθαρο το μήπως τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη όλοι από κοινού θα πρέπει να βοηθήσουν να βρεθεί μία λύση, να καταλήξουμε σε κάποια αποτελεσματική στρατηγική που θα έχει στόχο την ένταξη και όχι την γετοποίηση των τσιγκάνων. Να μην έχουμε ένα καινούριο σιδηρούν παραπέτασμα. Να γίνει κοινωνική έκταση και κριτήριο βασικό να είναι ε, το δικαίωμα διαμονής ή παραμονής και όχι η ηθαγένεια. Γίνεται να το πετύχουμε αυτό σε σχέση με την αγαστή συνεργασία που θα πρέπει να αναπτύξουμε. Μιλήσατε για ορθές πρακτικές και άρα αυτό θα πρέπει να το μεταλαμπαδεύσετε παντού ανάλογα με το που έχει επιτυχώς εφαρμοστεί. Πρώτα. ευχαριστώ πολύ. Επίτροπη. Συμφωνώ με όλους αυτούς οι οποίοι είπαν ότι απαιτείται να επενδύσουμε πράγματι στα παιδιά και στους ανηλίκους γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό και των προτάσεων τις οποίες έχει κάνει η συγχυτριά σας. Αυτή είναι και η βασική δική μας προτεραιότητα για το πρόγραμμα δράσης. Πρόγραμμα δράσης το οποίο θα προέλθει από την Task Force και τις προτάσεις της αλλά φυσικά απαιτείται μέχρι τότε η Task Force αυτή να αναλύσει προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια τα οποία ήταν διαθέσιμα ή και τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δαπανηθεί όταν έχει υπάρξει και τέτοιο φαινόμενο. Και τι θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε με ρεαλιστικό τρόπο να προχωρήσουμε σωστά και να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και επίσης και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τώρα για τη χάρτα. Η χάρτα είναι κάτι το σχετικά νέο. Οι επιπτώσεις της ύπαρξης της χάρτας στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι κάτι το οποίο έχει, θα έλεγα, ενσωματωθεί πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα σταδιακά. Τον Οκτώβριο θα παρουσιάσω μια ανάλυση του τι θα αλλάξει η χάρτα αυτή για τις νομοθετικές δραστηριότητες και την εφαρμογή των νόμων σε εθνικό επίπεδο. Και φυσικά θα έρθω και στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσω την, μελέτη αυτή. Υπήρξαν κάποιες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για το γιατί η οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση, μια οδηγία του 2004, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Γαλλία είναι μια τέτοια περίπτωση γιατί δεν έχει εφαρμοστεί και γιατί δεν έχουμε αντιδράσει τόσο καιρό. Εγώ θα ήθελα να σας επαναλάβω αυτό το οποίο είπα κατά τη διάρκεια της ακροάσεως που έκανα είχα πει ότι στον τομέα των ελευθεριών είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση τώρα όπου έχουμε στη διάθεσή μας τη χάρτα από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε μια νέα διάσταση και θα πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών. Όχι μόνο τις συγκεκριμένες οδηγίες. υπάρχουν και άλλες οι οποίες δεν έχουν πλήρως εφαρμοστεί. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω αμέσως να βλέπω το τι συμβαίνει στις χώρες μέλη και να συνεργάζομαι με τις χώρες μέλη έτσι ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι να παραπέμψουμε τα κράτη-μέλη στο δικαστήριο, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Το θέμα είναι να αλλάξει η κατάσταση στη βάση, σε επίπεδο πληθυσμού, σε επίπεδο πολιτών και αυτό ξεκίνησα να κάνω τον μήνα Φεβρουάριο επί τη βάση της οδηγίας 2004. Υπάρχουν κρατημέλη τα οποία έχουν κάνει θετικά βήματα. Υπάρχουν κρατημέλη τα οποία επιλύουν τα προβλήματα που υπάρχουν στις νομοθετικές τους διατάξεις και στις εφαρμοστικές τους διατάξεις. Υπάρχουν κρατημέλη με τα οποία έχω δυσκολία σχετικά με τις κινήσεις τους και υπάρχουν και άλλα κρατημέλη τα οποία δεν κινούνται καθόλου. Λοιπόν, έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία μπροστά μας. Εάν τα διαδικαστικά αυτά δικαιώματα είχαν εφαρμοστεί πλήρως και είχαν ενσωματωθεί στη γαλλική νομοθεσία, δεν θα υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία είδαμε κατά τη διάρκεια του θέρους. Συνεπώς λοιπόν τα διαδικαστικά αυτά δικαιώματα συνδέονται με την Οδηγία 2004 και με τις μορφές διακρίσεως οι οποίες συνέβησαν ή μπορεί να συνέβησαν εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Τώρα τι θα κάνουμε αν δεν απαντήσουν οι γαλλικές αρχές. Καλή ερώτησή σας. Εγώ υπολογίζω στις γαλλικές αρχές. Νομίζω ότι οι γαλλικές αρχές στο υψηλότατο επίπεδο της γαλλικής διοίκησης είπαν ότι θα ανταποκριθούν πλήρως και θα δώσουν απαντήσεις ε, ε, στις ερωτήσεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα της συνθήκη τους θέτει. Και αυτό θα λύσει τα προβλήματα. Ήδη μπορέσαμε μέσω των παρεμβάσεών μας να αλλάξουμε την εγκύκλιο την Υπουργική της 5ης Οκτωβρίου η οποία παραβίαζε κάθε σε ευρωπαϊκή ρύθμιση που μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ λοιπόν εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ρώτησα τις γαλλικές αρχές πώς εφαρμόστηκε η νέα εγκύκλειος. Ποια είναι τα δικαιώματα των μεμονωμένων πολιτών γιατί εδώ δεν μιλάμε για τα δικαιώματα μόνο μιας ομάδας, αλλά των μεμονωμένων πολιτών. Τα διαδικαστικά δικαιώματα, σαν παράδειγμα, έχουν τύχη εγγυήσεων προς αυτούς τους πολίτες, ναι ή όχι. Και αν έχουν τύχη εγγυήσεων, πού είναι οι αποδείξεις και θα πρέπει να έχω βρεθικά τα στοιχεία. Λοιπόν, περιμένω τα στοιχεία αυτά, θα αναλύσω τις απαντήσεις με την νομική μας υπηρεσία η οποία σαφώς είπε ότι απαιτούνται οι ερωτήσεις αυτές πριν προχωρήσουμε στην διαδικασία επιπαραβάση ή παραλήψη. Ας δώσουμε λοιπόν στην Γαλλία την δυνατότητα να απαντήσει πλήρως και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που θέτουμε. Ο Ετέρος Επίτροπος, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στη Φιλανδία για μια ακόμη φορά. Είχα πάει εκεί το Μάιο και σε μια συνάντηση με την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τον τύπο το βασικό θέμα ήταν η Ρωμά. Ήταν υπερήφανη για την ενσωμάτωση του τοπικού πληθυσμού των Ρωμά και δεν μπορούσαν να καταλάβουν το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες μέλη. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, να δούμε τι εμπειρίες έχουμε σε τέτοιες χώρες. Φυσικά το περιβάλλον και οι συνθήκες είναι διαφορετικές Παρ' όλα αυτά έχουμε πολλά να μάθουμε από τους Φιλανδούς και από αυτούς οι οποίοι έχουν θα έλεγα πείρα σε επίπεδο θετικών δράσεων, σε επίπεδο στοχευμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε επίπεδο παρεμβάσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όχι μόνο σε υψηλή ειδίκευση ε, θέσεις εργασίας αλλά και σε, χαμηλότερης, ε, σε χαμηλότερο επίπεδο θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή που κάνουμε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα βήματα για την καταπολέμηση της ένδυας και της υποαπασχόλησης είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν σε σχέση με τους Ρωμά, το θέμα της, ε, των μικροπιστώσεων επίσης, των πιστοτικών δηλαδή μικρού μεγέθους παρεμβάσεων, είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε σε χώρες όπως στα Ανατολικά Βαλκάνια. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, το θέμα είναι και κοινωνικό επαναλαμβάνω, θίγονται μικρές ή μεγαλύτερες κοινότητες, και οι κοινότητες αυτές ε, μπορούν εφόσον στέκονται καλά στα πόδια τους να προστατεύσουν τα μέλη τους από τον αποκλεισμό τον κοινωνικό. Είχα μιλήσει και με εκπροσώπους της Καθολικής Εκκλησίας σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που ο ρόλος των εκκλησιών είναι σημαντικός μερικές φορές στους πληθυσμούς των Ρωμά θα συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές και οι εκκλησίες. Θα συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκομένους, μεταξύ των οποίων και τις εκκλησίες, αλλά να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι θα υπάρξει μια μαγική λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο χαίνει εδώ και δεκαετίες θα έλεγα. Ακόμα και αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ακόμα και αν βρούμε τα καλύτερα δυνατά προγράμματα, σίγουρα θα υπάρξει, θα χρειαστεί χρόνος. Λοιπόν, δεύτερος γύρος. Κυρία Φιγουερέδο από την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι οι ενέργειες της Γαλλίας και άλλων χωρών ίσως εις βάρος των Ρωμά προκάλεσαν το ενδιαφέρον. Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις και από πλευράς νομικής. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ένα πράγμα εδώ. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτά τα οποία είπε η Επίτροπος Ρέντινγκ εδώ και λίγα λεπτά. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε απλά να λέμε λόγια καλά. Τα λόγια δεν αρκούν. Απαιτούνται δράσεις. Και για να αναλάβουμε δράσεις θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας συνολικές πολιτικές που να περιλαμβάνουν την απασχόληση, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την καταπολέμηση της ανεργίας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες ε, να ε, βλέπουν ότι τα προβλήματά τους την χάνουν αντιμετώπισης και να μην χρησιμοποιούνται οι Ρωμά μόνο και μόνο σαν μέσο αποτροπής από το να ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα. Το θέμα είναι επίσης όχι μόνο το οικονομικό αλλά και το πολιτιστικό και κοινωνικό. σε ένα λεπτό. Το ότι αυτοί οι οποίοι διώχθηκαν, ήταν Ρωμά, ε, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι διώχθηκαν επειδή ήταν Ρωμά. Νομίζω ότι πολλοί πιστεύουν σε κάποιες γενικεύσεις οι οποίες θα πρέπει να αποφευχθούν από μία στιγμή και μετά. Παρά βέβαια και την στάση του ηγέτη της σοσιαλιστικής ομάδας, ο οποίος χαρακτήρισε τους Ρωμά σαν μια δύσκολη μειονότητα, εμείς ε, είπαμε ότι υπάρχει ανάγκη και για την ε, παρακολούθηση της εφαρμογής του ποινικού κώδικα. Η Ρωμά όχι καθολικά, όχι γενικά, αλλά δυσανάλογα ε, σε μεγάλο ποσοστό ασχολούνται με παράνομες ενέργειες. Είχα θέσει μια ερώτηση σε σχέση με αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούνται, ε, αν υπάρχουν μειονότητες που εκπροσωπούνται σε κάποιες δραστηριότητες όπως ε, η εμπορία λευκής σαρκός ε, και σε επίπεδο φυσικά εκμεταλλευτών και εκμεταλλευομένων και η Ιντερπολ απάντησε ότι οι Ρωμά ανήκουν και στις δύο αυτές κατηγορίες. Η κυρία Μπλινκεβισίουτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα με τους Ρωμά έξι, την αποτυχία της γαλλικής κυβέρνησης να ενσωματώσει στο ιστορικό δίκαιο την κοινοτική οδηγία. Κατόπιν ξέσπασε ε, ένα γενικότερο σκάνδαλο και για άλλη μέρη τα οποία δεν μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο με τη Γαλλία. Άρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εξωθήσει τα κράτη-μέλη σε συμμόρφωση. και εκταμιεύονται συνέχεια χρήματα για την κοινωνική πλαισίωση των ε, Ρωμά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Όλο λόγια είμαστε εδώ. Γιατί δεν έχουμε πετύχει το συγκεκριμένο. μήπω θα έπρεπε να ξεκινήσει μια εκστρατεία συνειδητοποίηση. Ο επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν είχα δέκα λεπτά στη διάθεσή μου θα απαντούσα στα περισσότερα που ρώτησαν οι συνάδελφοι σε σχέση με το πρόβλημα που έχουμε στην χώρα μου, στην ε, Ρουμανία. Έχω υλικό, έχω τεκμηρίωση που θα μπορούσα να το θέσω στη διάθεση των ε, επιτρόπων. Όντως είναι μεγάλες δυσκολίες, μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε. Ήλχε ότι ποτέ δεν εντοπίστηκε σε όλου τι πραγματικέ διαστάσει το πρόβλημα των ε, τσιγκάρων. Γιατί το πρόβλημα πάντα ήταν ότι δεν υπάρχει ένα και μόνο κράτος το οποίο να συνδεθεί με την εθνότητα των ε, τσιγκάνων. Όντω έχουν πολλέ πτυχέ στο θέμα, γι' αυτό και θεωρούμε ότι έχει δίκιο η Κομισιόν. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια σειρά κινήσεων και μια αγωγή επί παραβάσεω, ούτω ώστε να σταματήσουν αυτά το οποία έγινε στη Γαλλία, αλλά επίση να είναι και αποτρεπτική αυτή η κίνηση σε όσου διανοούνται να κάνουν όσα έκανε η Γαλλία. Θα πρέπει επομένω να έχει μια ε, κοινοτική, πανενωσιακή πολιτική η Κομισιόν. Ο επόμενο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, θα μιλήσω μόνο ένα λεπτό γιατί έχει οριστεί ο κύριος Κολίνο ως ε, συντονιστής. Πρόβλημα δεν γίνονται μόνο τέτοια πράγματα με τους Τσικάνους ε, αλλά και με άλλους Ευρωπαίους. Πολλοί έχουν υποστεί συλλογικές κυρώσεις γιατί χρησιμοποίησαν την μητρική τους γλώσσα και μόνο. Οπότε έχουν παραβεί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αντιδρούμε αποφασιστικά, γιατί δυστυχώ υπάρχουν κράτη-μέλη όπου δεν υπάρχουν προβλήματα με εθνότητες, δεν υπάρχουν προβλήματα με τους Τσιγκάνους, διότι αυτό το κράτος αρνείται την ύπαρξη των προβλημάτων και των μειονοτήτων. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει καταστολή εκ των υστέρων, αλλά το πιο σωστό θα είναι να, να, να, προλαμβάνουμε αυτά τα προβλήματα. Μην διανοείται κάποιο κράτο μέλος να κάνει τέτοια πράγματα. κυρία Μποσκιούρτ θα απαντήσει αντί για μένα σε ερωτήσει τη κυρίας ε, Ρέντιν. Ναι κυρία Ρέντιν. Θα ήθελα περαιτέρω διευκρινήσει επί όσων είπατε, λέει κύριε είπατε για περιπτωσιακή εξέταση, περιπτωσιολογική εξέταση των όσων έχουν γίνει αυτών των ε, απελάσεων. Όμως, έγιναν και ομαδικές. Άργησε η εγκύκλειος να διορθωθεί και γι' αυτό επί τη βάση της εθνοτικής τους καταγωγής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκδιώχθηκαν από τη Γαλλία. Εσείς θα κάνετε να εξετάσετε την κάθε περίπτωση χωριστά. Για κοιτάξτε αυτήν την εγκύκλιο. Τα πράγματα εκεί είναι ξεκάθαρα. Το, το, το, το τι έγινε και φυσικά πρόκειται περιορισμένο διάκριση. Ο επόμενο. Θα ήθελα να πω τα εξή. Δύο θέματα αρχέ. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία βελτιώνει τους όρους ε, διαβίωσης των Ρωμά και ταυτόχρονα βελτιώνει την εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι η πρώτη φορά αυτή κατά την οποία η Κομισιόν ε, παίζει το ρόλο του ελεγκτή. Ελέγχει δηλαδή την εφαρμογή των ε, βασικών δικαιωμάτων. Για πρώτη φορά εδώ έχουμε μία υπόθεση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τέτοιο τρόπο. Και σωστά αναφερθήκατε στη Φιλανδία, γιατί στη Φιλανδία αναρωτιέται κανένας πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσοι, τόσοι ζητιάνοι σε μια χώρα που χρειάζεται να απελευθούν τα Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν. Και ενθουσιάστηκα από τη δυναμική παρέμβασή σα. Σήμερα ξανά έχετε αναφερθεί στο, στην ανάγκη σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων για του Ρωμά. Εγώ θα προσθέσω και για άλλου, ε, γιατί υπάρχουν πολλέ μειονότητε και άλλοι που υποφέρουν και δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Επειδή είμαι από την Κύπρο και γνωρίζω ότι πολλές φορές ακούσαμε για το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δημοκρατικά ελλείμματα και δεν υπάρχουν μηχανισμοί πρακτικής υλοποίησης ευρωπαϊκών οδηγιών, ευρωπαϊκών ψηφισμάτων, της ίδιας της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διαρωτούμε από πού αντλείται αυτό το πείσμα, την ελπίδα και τη δύναμη ότι τώρα με αφορμή του Ρωμά θα υπάρχουν εκείνοι πρακτικοί τρόποι υλοποίηση των όσων λέτε. Θα ήθελα πραγματικά έμπρακτα να δω ότι όλα αυτά τα οποία λέμε δεν είναι απλά λόγια και διακηρύξεις αλλά θα υλοποιηθούν στην πράξη. διαφορετικά θα αμφισβητήσω γιατί 36 χρόνια περιμένουμε δικαιοσύνη και δεν την έχουμε στη χώρα μου. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ευχαριστώ που την επόμενη άνοιξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Ρέντι συγκεκριμένη, θα ζητήσει συγκεκριμένες ε, ε, πληροφορίες για το πώς θα πανούν τα χρήματα από τα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Πα, εκ παραλίλου τα εν λόγω κράτη-μέλη να δώσουν πραγματικές πληροφορίες όσον αφορά τις δομές μέσω των οποίων έχουν δράσει στα περασμένα χρόνια γιατί σε χώρες όπως η Βουλγαρία παραδείγματο χάρη, πολύ σημαντικά σημαντικές οντότητες που ήταν στο παρελθόν σημαντικές στον τομέα της ώρα, των Ρωμά, εξαφανίστηκαν. Γιατί η Επιτροπή κατά των διακρίσεων στη χώρα μου έχει μειωθεί όσον αφορά το μέγεθός τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά όργανα που εξαφανίζονται αντί να δυναμωθούν για να λειτουργήσουν καλύτερα. <clears throat> δηλαδή, μόνο το αριθμό πόσα χρήματα δαπανήθηκαν δεν θα μας δώσει επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Gostava Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σας στηρίζουμε 100%. Είναι κοινή μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί πρόκειται εδώ για κάποιους Ευρωπαίους πολίτες και στην χώρα μου. Με επιτυχία έχουμε ένα πρόγραμμα με κονδύλια ευρωπαϊκά. Πρόγραμμα πάρα πολύ πετυχημένο για τους ε, τσιγκάνους. Αλλά έχει αναφερθεί ότι πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το να υπάρχει πολιτική βούληση και πολιτική πυγμή πλευρά πολιτικής ηγεσία για να προχωρήσουμε στην ένταξη, την κοινωνική των συγκάνων. Είχαμε παράγοντες δηλώσεις εκ μέρους των Ρουμανικών Αρχών για τις δυσκολίες που έχουν όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των τσιγκανών ε, στην χώρα εκείνη. Ε, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν προκαταλήψεις. Well, President, I Η Επίτροπη πάλι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιταχθούμε, να μην πνιγούμε εδώ, να μην καταποντιστούμε. Άσχετα αν πρόκειται για μικρή ή μεγάλη χώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιταχθεί και θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της. Για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει να έχουμε μια πολύ σαφή νομική υπόθεση. Και γι' αυτό το Φεβρουάριο του 2011 θα αρχίσουμε να εξετάζουμε όλα τα κράτη-μέλη σχετικά με την εφαρμογή, τη μη εφαρμογή της οδηγίας ελεύθερης διακίνησης. Γιατί αυτή δεν είναι μία τυχαία ε, οδηγία μαζί με όλες τις άλλες πρόκειται για μια οδηγία που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μειώνει τις δυνατότητες ενός κράτους να δράσει κατά εκείνων των ατόμων που δρούν εγκληματικά. Τουναντίον η οδηγία ορίζει τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη είτε ε, όταν υπάρχουν λιγότεροι από τρεις μήνες ή περισσότερο από τρεις μήνες διαμονή σε μια χώρα. Αλλά κάθε ένα άτομο, κάθε ένας Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται βάσει δικοσικών κανόνων που τον προστατεύουν ακόμα και αν κατηγορείται για παραπτώματα και θα πρέπει να φροντίσουμε αυτοί οι κανόνες όλοι να εφαρμοστούν και διασυνοριακά. Και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουμε εδώ επιτάπτως είναι να πραγματοποιήσουμε την ύπερο της δικαιοσύνης και να μην έχουμε ε, διακρίσει κατά κάποιων ομάδων πολιτών. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα νέο περιβάλλον γιατί έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας που εφαρμόζεται και στον τομέα της δικαιοσύνης και γιατί έχουμε την Χάρτα Βασικών Δικαιωμάτων η οποία επίσης εφαρμ... ισχύει για όλα τα επίπεδα και θα πρέπει εσείς ως κοινοβούλιο, εμείς ως Κομισιό θα πρέπει να ε, υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα αυτά. Λέγεται ότι καταψήφισε, δεν ακολούθησε, δεν δίωξε η Κομισιόν. Όχι του εναντίον, για πρώτη φορά έχει ξεκινήσει σαν σύνολο μία επιπαραβάση διαδικασία και το δήλωσε αυτό σαφώς μεγαλόφωνα και δημόσια. Μην υποτιμάτε λοιπόν την ε, ισχύ των δράσεων αυτών της Κομισιόν σήμερα. Δεν είναι και απόλυτη δράση, γιατί η Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει κάποιους κανόνες δεν μπορεί να κάνει κάτι επειδή κάποια ιδέα της πέρασε και να πει αυτό εκείνο θα γίνει. Όχι, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες. Είδαμε τη δυνατότητα εφαρμογή τη οδηγία, έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε και δράσαμε. Εάν εντωμεταξύ το πρόβλημα επιληθεί ή αν επιληθεί για κάποιο άλλο κράτο μέρο, δεν χρειάζεται να περάσουμε στη διαδικασία την δικαστική. Όχι. Ξεκινήσαμε μια πολύ μακρά και χρονοβόρα διαδικασία και ελπίζω ειλικρινά ότι αυτές οι διαδικασίες που θα αρχίσουν σήμερα ή που θα αρχίσουν αύριο δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος αλλά σε ένα-δύο μήνες τα κράτη-μέλη θα έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Αυτό είναι που θα πρέπει να πετύχουμε. Τώρα, όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων, θα πρέπει πραγματικά να διευκολύσουμε τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε λεπτομέρειες, όχι για τη θεωρία, αλλά με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και άλλα στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά των αρχών σε σχέση με κάποιους μεμονωμένους πολίτες. <coughs> και χρειαζόμαστε έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμπεριφορά αυτή ή που αποδεικνύουν ότι όλα πήγαν καλά. Είναι όμως σημαντικό για μας να μην δεχθούμε γενικές πολιτικές διαβεβαιώσεις. Ας λάβετε υπόψη λοιπόν αυτό το σημαντικό βήμα προς τα εμπρός Και α έχει την υπόψη μα ότι είμαστε μια εκκληστική επιτροπή που εφαρμόζει αυτό που υπάρχει στι νέε συνθήκε. Δεν το έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο γιατί δεν το είχαμε πριν από τι συνθήκε αυτέ, δεν το είχαμε πριν από την κάρτα. Άλλαξε λοιπόν όλο το περιβάλλον και η αλλαγή αυτή του περιβάλλοντο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο εάν όλα τα θεσμικά όργανα κινούνται προ την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Επίτροπο Σάντερ να προσθέσω ίσως κάποιες διαστάσεις στη συζήτηση μέχρι τώρα. Υπάρχει ο λόγος γιατί το συζητάμε το θέμα αυτό μετά τα γεγονότα δηλαδή στη Γαλλία και την αντίδραση της Επιτροπής. Τα προβλήματα υπήρχαν από πριν. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έστρεφαν την προσοχή τους στο θέμα των Ρωμά. γιατί έβλεπαν τους Ρωμάς της να είναι άτακτοι θα έλεγα στις, στους δρόμους των πόλεων τους, δεν το ήξεραν αυτό στο παρελθόν και έμεναν εκτός της κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής λόγω ακριβών, ακριβώς και της οικονομικής κρίσης. να πω ότι στα διάφορα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά Ρωμά, φτάνω στο 8 με 10% του πληθυσμού, οι δημογραφικές τάσεις είναι σαφείς. Και βλέπουμε τώρα και τις επεδόσεις των σχολείων να κατεβαίνουν λόγω ακριβώς της αποτυχημένης συμπερίληψης, αν θέλετε, ενσωμάτωσης των Ρωμά και το ίδιο ισχύει και για την αγορά εργασίας, γιατί σε κάποιες περιοχές οι Ρωμά αντιπροσωπεύουν το 14% των νεοεισερχομένων στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν απώλειες λόγω ακριβώς του κοινωνικού αποκλεισμού και οι απώλειες αυτές είναι και οικονομικές και κοινωνικές και ηθικές αλλά επαναλαμβάνω και οικονομικές. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει λόγος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με συνολικό τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κοινωνικό ταμείο με αποτελεσματικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε σωστά και το Διαφθορτικό Ταμείο για να αναστρέψουμε τις τάσεις αυτές. Εγώ δεν φοβάμαι ότι θα χαθεί η όθηση η οποία υπάρχει σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει έρθει στο κέντρο της προσοχής και τα κοινωνικά αυτά προβλήματα παραμένουν μιας και η οικονομική κρίση συνεχίζεται και λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης υπάρχουν και οι κοινωνικές συνέπειες. Μίλησα με εκπροσώπους επίσης και της Ουγγρικής κυβέρνησης που θα ακολουθήσει τη Βελγική στην Προεδρία του Συμβουλίου και σκοπεύουν και αυτοί να κάνουν νέες προτάσεις για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια καλή συνεργασία. Προτείνουμε επίσης και ορισμένες πολιτιστικές παρεμβάσεις. Συζητήσαμε μέλη του Κοινοβουλίου να δείξουμε μία ταινία για τον τρόπο που ζουν οι Ρωμά στην Βόρεια Ουγγαρία. Αυτό θα εντυπωσιάσει όσους έχουν χρόνο να το δουν. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει υπάρξει μόνο πρόοδος ε, σε επίπεδο διοικητικό. Η βουλγαρική περίπτωση που είχε τεθεί είναι χαρακτηριστική. Υπάρχουν πολλά να μείνουν, να γίνουν εκεί. Υπάρχει ένα θέμα και στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου και των παρεμβάσεών του. Κάποιοι από αυτούς που εκπαιδεύτηκαν με τα χρήματα του Κοινωνικού Ταμείου αναγκαστήκαμε να τους απολύσουμε. Εγώ συναντήθηκα με τον Αντιπρόεδρο της Βουλγαρικής Κυβέρνησης προχθές και ήταν μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για τις βλέψεις της νέας κυβέρνησης και να του εξηγήσω και τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα με η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε την δυνατό, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα εις βάθος με την ρουμανική ε, κυβέρνηση σε υψηλότατο επίπεδο, ίσως και με τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο και εκπροσώπους της κυβέρνησης. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ένας διάλογος ο οποίος έχει προχωρήσει αρκετά και είμαι πεπισμένος ότι θα σημειωθούν βήματα προόδου. Ευχαριστώ. Τρίτος γύρος. Κλάες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ρέντινγκ αν ζητήσατε συγνώμη από τη γαλλική κυβέρνηση γιατί κάνατε μια γελία παρομοίωση με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, ε, τι ακριβώς έχει γίνει. Θα ήθελα να μάθω επίσης αν ξεκινάτε τέτοιες διαδικασίες και εις βάρος άλλων κρατών μελών. Πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνεται εδώ και λίγες εβδομάδες ότι θα υπάρξει έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία προορίζονται προς τους Ρωμά έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Τα προβλήματα το 2007 υπάρχουν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Και οι χώρες αυτές στην ουσία έχουν την τάση να εξάγουν τα προβλήματά τους σε άλλες χώρες μέλη εις βάρος των χωρών ε, στις οποίες καταλήγουν οι πληθυσμοί αυτοί. Πρέπει λοιπόν να υπευθυνοποιηθεί και η κοινότητα των Ρωμά. Ξέρετε ότι υπάρχει δυσανάλογη εγκληματικότητα από πλευράς των Ρωμά σε ορισμένες χώρες. Ε, χρησιμοποιούνται τα παιδιά για ζητιάνη κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τη Γαλλία, αφορά την Ευρώπη και η απάντηση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Το να επιτίθεται κανείς στη Γαλλία δεν λύνει το πρόβλημα της ουσίας. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η σωστή απάντηση, είναι κάτι το άδικο. Η Γαλλία είναι μια χώρα υποδοχής ε, πληθυσμών και ενσωματώνει πληθυσμούς από όλες τις περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί τίθεται το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη κοινότητα. Νομίζω ότι αυτοί που υποδέχονται τους πληθυσμούς των Ρωμά έχουν το δικαίωμα να τους βοηθούν να ενσωματωθούν, αλλά θα πρέπει και οι πληθυσμοί αυτοί να θελήσουν να ενσωματωθούν. Το να λέμε ότι η Γαλλία είναι ρατσιστική, ξενοφοβική κτλ. είναι εντελώς αδικό. Και ταυτόχρονα σε νομικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γιατί δεν έχουν υπάρξει σωστές λύσεις. Λοιπόν, το δικαίωμα στη διακίνηση την ελεύθερη είναι βασικό, αλλά θυμίζω ότι και τα παιδιά έχουν δικαιώματα να πάνε στο σχολείο, και δεν θα πρέπει να επιλέγεται η ζητιανιά σαν, σαν στυλ ζωής θα έλεγα. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ελαστικοί στις κρίσεις μας και δεν θα πρέπει ε, τέτοιες καταστάσεις να διονίζονται. Η απόφαση λοιπόν την οποία πήρατε είναι τέτοια που αν τυχόν σήμερα δεν βρει απάντηση τότε στην ουσία θα προχωρήσουμε σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Η κυρία Βερζά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω όπως άλλοι για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε την κατάσταση. Εγώ είμαι μεταξύ εκείνων των αλληλών που ανήχησαν με κάποιες δηλώσεις της γαλλικής κυβέρνησης και όχι επειδή το, η γαλλική κυβέρνηση κάνει κάποιες δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία ε, εξάπτεται. Κάποιοι ναι, αλλά όχι την πλειοψηφία των Γάλλων. Εγώ θεωρώ ότι δεν προχωράτε αρκετά γλυγορά, δεν σας εκπλήττει αυτό φαντάζομαι. Ε, μιλήσαμε πολύ για την εγκύκλωση της 5ης Αυγούστου η οποία αποσύρθηκε όπως και κάποια άλλη εκείνη της Ιουνίου. Από την άλλη μεριά, 9 ε, Αυγούστου, αλλά εκείνη τη 24 Ιουνίου δεν απεσύρθηκε. Με αυτή τη βάση συνεχίζονται οι απελάσει. Με αυτή τη βάση συνεχίζεται ε, η κατάσταση να επιδεινώνεται στην κατάσταση και νομίζω ότι και η εγκύκλειος ε, και η εγκύκλωση 24 Ιουνίου λέει να απελάσσονται ε, οι νομάρχοι, ε, να οι άτομα που ε, κάνουν διάφορα παραπτώματα που αναφέρονται εκεί. Η εγκύκλωση αυτή ζητάει από τους νομάρχες και τους επάρχους να πάρει μέτρα απομάκρυνσης ε, εκείνων που βρίσκονται σε αυτά τα στρατόπεδα αν δεν έχουν τη γαλλική υπηκότητα. Ναι, παιδιά, ξέρουμε ότι οι απελάσεις αυτέ γίνονται συστηματικά και άμεσα όταν πρόκειται για Ρωμά. Θέλετε αποδεικτικά στοιχεία? Εάν ναι, κύριε ε, Ρέντινγκ, εγώ θα κάνω σήμερα μια επίσημη έκκληση σε όλου του δημάρχους να σας αποστείλουν αυτά τα στοιχεία. Τελειώνω, τελειώνω, πρόεδρο. Η εγκύκλωση στις 13 Σεπτεμβρίου αναφέρεται σε 441 άτομα που ε, απελέσταν. Νομίζω ότι η γαλλική κυβέρνηση θα μπορούσε να σας αναφέρει στον κατάλογο αυτών των ομάδων και στα ονόματα των ατόμων αυτών. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σας ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, για την καθυστέρηση. Ο κ. Παντρεστόκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο όμω. Ε, κυρία Ρέντινγκ, ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία επί παραβάση κατά της Γαλλίας. Από την άλλη μεριά όμως η Γαλλία νομίζω ότι τηρεί την νομοθεσία. Ζητάτε τότε από τη γαλλική κυβέρνηση να τροποποιήσει την νομοθεσία της. εάν, έχετε, εάν υπάρχουν κάποιες ε, ε, κάποια προβλήματα, αν έχουν Γάλλοι υπήκοοι κάποια προβλήματα, μπορούν από μόνοι τους να προσφέρουν κατά της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται για θέματα της Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να ερμηνεύσουν τα, ε, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό. Πρόκειται για θέματα ανεξαρτησίας. Είναι σαφέστατο. Εγώ θα ζητούσα να υπάρχει μια ανεξάρτητη έρευνα γιατί αυτά που δεν ήρθαν βέβαια είναι φοβερά αλλά από την άλλη μεριά ακόμα φρικτότερο να υπάρχει εκ των έξω παρέμβαση θα ήθελα να εξετάσει η πιο εις βάθος τα πράγματα αυτά κύριε Ρέντινγκ uh, Νομίζω ότι λείπει εδώ η, η πτυχή της ισότητας των φίλων. Να έρθουν από εδώ πέρα οι γυναίκες, οι τσιγκάρες για να μας πούνε τι γίνεται εδώ πέρα με τη μαζική με παρέμβαση των δημιουργικών τους και με αυτή τη μαζική δυσμενή ε, διάκριση την οποία εφίστανται μέσα στην ίδια τους την κοινότητα. Για όλα αυτά τα παιδάκια που δεν τα αφήνουν να πάνε σχολείο. Θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, να κάνουν οικοκυριό και αναγκάζονται να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις και να, να, να, να, να γεννάνε. Να, τι γίνεται με την κοινωνική ένταξη. Θέλω να ακούσω τις μαρτυρίες, καταθέσεις για αυτού του είδους, τον εμπόριο λευκή σαρκός, την εκπόρνευση, όλα αυτά που υφίστανται γιατί η σύγχρονη θεωρία δικαιωμάτων λέει ότι κατά τον ιδιωτικό βίο η παραβίαση των δικαιωμάτων θα πρέπει να σαν έγκλημα από ένα κράτος και επομένω, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση θετική κατά αυτών των μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μην ξεχνούμε, Πρόεδρε, ότι μιλούμε εδώ για κάποιους οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει παράνομα στο έδαφος που ανήκει σε κάποιον άλλο και ε, τους διώχνουν διότι έχουν παρανομήσει και είναι άνεργοι γιατί δεν ψάχνουν καν δουλειά και όχι μόνο στη Γαλλία και στη δική μου την περιφέρεια έχουμε σημαντικά προβλήματα με τέτοιου είδους ε, ε, στρατόπεδα, συνοικισμούς, εγκαταστάσεις. Τι γίνεται, όλοι λένε εδώ πέρα για τα δικαιώματα κατά των, δικαι... των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παραδίασή τους δηλαδή, και κανείς δεν λέει για το δικαίωμα όμως στην ε, ιδιοκτησία, για τις ζημίες που προξενούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που κατασκηνώνουν και η κυρία Ρεντίν θέλει να τους προστατεύσει τους τσιγκάνους. Μα τι γίνεται, θέλετε να προστατεύσει και το δικαίωμα του να κατασκηνώνει κανείς παράνομα στο ακίνητο κάποιο άλλο, φυσικά και έχουν δικαίωμα. Αλλά έχει και υπόλοιπη κοινωνία και όλοι μας έχουμε. Και αυτοί που είναι οι κύριοι του ακινήτου που κατασκηνώνουν οι Τζιγκάνοι. Και αυτοί που θέλουν να του εντάξουν κοινωνικά, ρώτησαν του Τζιγκάνους, θέλουν να ενταχθούν, θέλουν να μείνουν σε εργατική πολυκατοικία, θέλουν να μείνουν κάπου μόνιμα. Μα το, το, το, το, το τρόπο ζωή του ακριβώ είναι νομαδικό και ακριβώ το πρόβλημα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για τη συνεργασία σα. Έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο για τι καταληκτικές παρατηρήσει των Επιτρόπων και πρώτη η κυρία Ρέντινγκ. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, το 80% αυτών των ανθρώπων που είναι στις λεγόμενες παράνομες κατασκηνώσεις έχουν την γαλλική ηθαγένεια. Έχουμε διατάξει εθνικού δικαίου, ευρωπαϊκών δικαίων που βεβαίω δίνουν ε, την ε, εξουσία σε ένα κράτος να ασκεί και δικαιοδοσία κατά το οποίο αφορά άτομα, φυσικά πρόσωπα και όχι ομάδες προσώπων. Και είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊκές οδικίες θα πρέπει να εφαρμόζονται, θα πρέπει να εντάσσονται στο ιστορικό δίκαιο και αυτό δεν είναι στην κριτική ευχαίρεια του κράτους, είναι μια υποχρέωση. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αντίστοιχα την επιλογή. Έχει την υποχρέωση να φροντίσει να πραγματοποιείται κάτι τέτοιο και αυτό είναι ο τρόπος για τον οποίο ε, έχει αποφασιστεί να ακολουθηθεί η αγωγή επί παραβιάση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτός είναι ο συνήθις τρόπος κατά τον οποίο λειτουργούν ε, θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Ότι η απόφαση σε σχέση με το τι είναι κοινωτικό δίκαιο και τι δεν είναι, δεν είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό κρίνεται από τους συννομοθέτες. Από το Συμβούλιο της Κυβερνήσης, από τους Υπουργούς, από όλα τα κράτη-μέλη, οι οποίοι έρχονται σε συνεννόηση και συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι γίνεται η νομοπαρασκευαστική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν συμφωνία κοινή των κρατών μελών, τα οποία οφείλουν μετά και να εφαρμόσουν αυτό το δίκαιο το οποίο θεσπίστηκε. Τα συμπεφωνημένα πρέπει να τηρούνται. Πάκτα σουν τη σερβάντα. Έτσι λειτουργεί εύρυθμα κάθε θεσμικό όργανο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάμβανε κάποια απόφαση μόνο επί τη βάση των κείμενων διατάξεων δηλαδή. Αυτό το πει και τώρα θα πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για τη Γαλλία. Και για άλλους. Ελπίζουμε δε ότι όλη αυτή η φασαρία εξυπηρέτησε. Βοήθησε, ωφέλησε σε κάτι. Τότε δηλαδή τώρα όλες οι κυβερνήσεις αισθάνονται ότι έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης της φτώχειας που δεν είναι μόνο πρόβλημα των τσιγκάνων. Θα πρέπει όλοι τώρα να, έχουν καταλάβει ότι όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν να μην υπάρχουν διακρίσεις κατά των γυναικών. Κάτι το οποίο σοβεί στην τσιγκάνικη κοινότητα και το ξέρουμε. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πλαισίωση των ανηλίκων από κάποια τρυφερή ηλικία και γι' αυτό τα παιδάκια των τσιγκάνων και ιδίω τα κοριτσάκια θα πρέπει να έχουν προσβασιμότητα στο σχολείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζω το θέμα αυτό από την Task Force που είπαμε που αναλύει τα κονδύλια που απορροφώνται ή ου. Και επομένως γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα αυτής της Task Force τα οποία συμπεράσματα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν κατά τα τέλη του νεστότος έτους. Άρα, επί τη βάση των συμπερασμάτων αυτών, τότε θα προχωρήσουμε. Και γι' αυτό και θεωρώ θετικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα. Και για το πώ θα συνεργαστούμε, ούτω ώστε αυτή η απάνθρωπη κατάσταση αυτών των μειονοτήτων των Ρωμά μπορούν στο μέλλον να βοηθηθούν. Συμφωνώ με όλου αυτού που ρεαλιστικά το αντιμετώπισαν και είπαν ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που σοβεί εδώ και αιώνε. Δεν μπορεί επομένω με μία απόφαση διαμαγείας να λυθεί. Μπορεί όμως να λυθεί όταν όλοι αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να γίνει αλλαγή στις νοοτροπίες και έτσι να προσπαθήσουμε να σώσουμε την επόμενη γενιά συγκάνων. Που τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι παιδιά και έτσι με μια διαφορετική νοοτροπία να μπορέσουμε να τους δώσουμε μια καλύτερη ζωή. Πέραν αυτών, όλα όσα συζητούμε εδώ έχουν ως βάση, κάθε συζήτηση έχει ως βάση τις συνθήκες που με τη σειρά τους εκπηγάζουν από την κοινή βούληση των Ευρωπαίων από τη δεκαετία του 50. Αποφασίσαμε έτσι να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον με πλατφόρμα τις κοινέ αξίες οι οποίες είναι η υψίστη προτεραιότητά μας. Δυστυχώς στο παρελθόν δεν επικαλεστήκαμε αρκετά αυτές τις αξίες γι' αυτό και ελπίζω ότι τώρα και στο εξής οι αξίες θα διέπουν την πολιτική μας δράση, την νομοπαρασκευαστική διαδικασία, την εφαρμογή των νόμων, την ατζέντα των δραστηριοτήτων μας. Αυτές οι αξίες θα έχουν την ύψιστη θέση. Αυτές αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι θέμα επιλογής διακριτικής ή είναι επιταγή για όλους. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας να μείνετε στα κεντρικά θέματα και να μας δώσετε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις τις σημαντικές που ακούσαμε εδώ. Επί Άντερ, Μία ερώτηση, η οποία θεωρώ ότι είναι κομβική οι Ρώμα θέλουν να ενσωματωθούν. Είναι σημαντικό να προσπαθήσει να, ερμηνεύσει, να καλά το τι εννοούμε με τη λέξη ενσωμάτωση και να προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα και από την πλευρά των Ρωμά. Εμείς δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση τη δημιουργία μιας ομοιογενούς ε, κοινωνίας και την κατάργηση της ποικιλότητα της κοινωνίας αυτής. Μιλάμε για μια κοινωνία με διαφορές, ποικιλόμορφη, αλλά όπου τα δικαιώματα θα είναι καθολικά. Η δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνία και σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες θα είναι ανοιχτή σε όλους. Είναι αλήθεια ότι στους τελευταίους αιώνες οι Ρωμά έζησαν στην Κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια στα όρια της κοινωνίας. Είναι επίσης αλήθεια ότι πριν από τις αλλαγές της δεκαετίας του 90 η πλειοψηφία των Ρωμά είχαν θέσεις απασχόλησης και ε, κατά κάποιο τρόπο ήταν ενσωματωμένοι στις κοινωνίες τους. Αν και ε, οι περισσότερες από τις θέσεις απασχόλησης που είχαν ε, δεν ήταν υψηλής εξειδίκευση. Αλλά δούλευαν και στη βαριά βιομηχανία και στις οικοδομές κτλ τις έχασαν αυτές τις θέσεις απασχόλησης και ήταν δυστυχής από αυτό το φαινόμενο. Και αυτό οδήγησε στην, στον αποκλεισμό τους από τις κοινωνικές δομές σε ορισμένες φτωχές περιοχές. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες είδαμε την εμφάνιση ορισμένων ιδιαίτερα περίπλοκων κοινωνικών προβλημάτων που οδήγησαν στην απόλυτη ένδια. Έλλειψη εκπαίδευσης, έλλειψη κατάρτισης, φυσικά αναλφαβητισμός, στέρηση δικαιωμάτων και από εκεί και πέρα ήταν ένα μικρό βήμα η παρανομία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να, κατανοητό, να γίνει κατανοητό είναι ότι μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας η οικονομική ύφεση καθιστά πάρα πολύ δύσκολη τη συμβίωση ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και δημιουργεί πολιτικές εντάσεις. Μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο. Θα πρέπει να σπάσει ο φαύλος αυτός κύκλος, θα πρέπει να αντιστραφούν οι τάσεις αυτές όσο δύσκολο και αν είναι και θα το πετύχουμε αυτό αν έχουμε κοινό τρόπο κατανόησης των προκλήσεων που μας περιμένουν. Ευχαριστώ το Πάντερ. Μια συνεδρίαση που κράτησε δυόμιση ώρες, ίσως να ήταν λίγο κουραστική, αλλά νομίζω ότι ήταν καρποφόρα. Υπήρξε ένταση στην ανταλλαγή απόψεων και τώρα θα ακούσουμε τις τελικές παρατηρήσεις από την πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης, την κυρία Μπερές, και μετά θα τερματιστούν οι εργασίες μας. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για αυτή την κοινή ακρόαση. Ήταν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να κάνει σήμερα τη συζήτηση αυτή. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει έχοντας ακούσει τους τρεις επιτρόπους είναι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα θέμα που άπτεται των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος είπε ότι έχουμε να κάνουμε με τη θέση σε ισχύ της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κάτι το οποίο αν μοίρασε ξανά τα χαρτιά και έχουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη βάση για μια αποτελεσματική δράση. Πόσο μάλλον που όπως βλέπουμε δεν έχουμε φύγει ακόμα από την κρίση. Στα πλαίσια της κρίσης αυτής, ό,τι μπορεί να προκαλέσει ε, αντιδράσεις ε, και ανακλαστικά λαϊκισμού και εξενοφοβίας ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν εδώ με ένα παράδειγμα σαφέστατο και σε σχέση με τις διακρίσεις και σε σχέση με την ένδια και θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε στην Επιτροπή μας την πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να αναλυθεί στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Αυτή η πρωτοβουλία, η πιλωτική για την καταπολέμηση της έμβιας, γιατί θυμίζω ότι για τους Ρωμά θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία η στρατηγική αυτή, για την οποία θα πρέπει να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα. Τέλος, όταν ξεκινήσετε τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού ταμείου, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής για την προτινόμενη στρατηγική και για την συνεκτικότητα με τους στόχους της καταπολέμησης της στόχιας. Η εμπειρία μας δίνει το μάθημα σύμφωνα με το οποίο μια σωστή δημόσια παρέμβαση προαπαιτεί διοικητικές ικανότητες και σωστές συνθήκες διαλόγου με το σύνολο των πρωταγωνιστών. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να γίνει και για μια χώρα σαν τη Ρουμανία αλλά και για τη Γαλλία ακόμα μια τέτοια προσπάθεια πρέπει να αναλυφθεί γιατί οι συνθήκες διαλόγου με το σύνολο της κοινωνίας δεν ήταν πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη συνεργασία τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βελγική Προεδρία και να ευχαριστήσω και τον χαιρόν τον εκπρόσωπο, υπεύθυνο μάλλον, της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Να θυμίσουμε σε όλους ότι μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και της Χάρτας, η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση για αξίες, είναι συζήτηση για αρχές και αυτές οι αρχές και αξίες υπογραμμίστηκαν. Είναι δεσμευτικές οι νομικές ρυθμίσεις για την προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πολιτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περισσότερο από ποτέ ο θεματοφύλακας αυτών των νέων αρχών και αξιών των ενσωματωμένων στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κάνει ό,τι μπορεί και θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμηθούν πλήρως οι διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενσωματωθούν αυτοί οι πληθυσμοί στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Μένουν πολλά να γίνουν, ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά έστω και λίγο συνεισφέραμε στις φιλοδοξίες αυτές, την πρωτοβουλία αυτή στα πλαίσια της συζήτησης και της συνάντησης που προηγήθηκε.